Right, good afternoon everybody. Um, well... Χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Νέα σύνοδο έχουμε τώρα μέχρι τις 5.30 και έχει έρθει η ώρα σήμερα του διαλόγου με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ, και προφανώς τον πρόεδρο της Ευρωζώνης, όπως βλέπετε τον πολύ γνωστό μας και εν ευθέτω χρόνο θα έρθει όλη η ΡΕΝ, Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ακολουθούν τα αποκρίσει και όπως σας είπα το πρωί, ε, αν θέλετε το λόγο να σηκώσετε τη ροζ κάρτα. Κανείς δεν μπερδεύτηκε το πρωί με τα χρώματα, μια χαρά τα πήγατε. Λοιπόν, Αρχίζουμε από τον πρόεδρευοντα του ΕΚΟΦΗΝ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ladies and gentlemen, uh, Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ στα αγγλικά ο Υπουργός, για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είμαστε μέσω της διαδικασίας διαλόγου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπροσωπώ εγώ ενώπιό σας σήμερα το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ που είναι το Συμβούλιο Υπουργών ε, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, γιατί και τα δύο έχουν σημασία και για την Επιτροπή σας. Και είμαστε ε, πολύ υπέρ ενός τριμερούς διαλόγου, σε στενή συνεργασία δηλαδή ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σάρων που μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε να σας συναντήσουμε. Θα ήθελα να σας πω αρχικά ότι σήμερα είναι η εθνική μας εορτή της Ουγγαρίας και αργία στην Ουγγαρία. Από ό,τι φαίνεται ο καιρός όμως είναι με το μέρο μας σήμερα, μας κάνει καλή μέρα. Άρχισε μια σειρά επαναστάσεων στο 19ο αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα συγκεκριμένα και στην Ουγγαρία έχουμε από τις πιο λαμπρές επαναστάσεις εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Ήταν η επανάσταση των αστών. Το 1848 ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου. Γι' αυτό ε, έχουμε σήμερα την επέτειο αυτής ε, της ιστορικής στιγμής για τη χώρα μας και μοναδική ευκαιρία ε, αυτή που έχω σήμερα να είμαι ενώπιόν σας. Um, ε, θα ήθελα συνεχίζοντας να σας πω ότι ε, θα πρέπει λίγο να σας περιγράψω το σκηνικό. Αυτό το καιρό η οικονομική διακυβέρνηση ε, κυριαρχεί και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Όπως, ε, όπως γνωρίζετε συμβαίνουν ε, τρομακτικά πράγματα, είναι φοβερές οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. Επίσης η εσωτερική ε, ζήτηση αρχίζει σιγά σιγά να ανακάμπτει και γενικότερα η ανάκαμψη φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης σίγουρα ε, δεν είναι παντού ίσος. Γι' αυτό έχουμε ανησυχίες που συνδέονται και με τη γεωπολιτική κατάσταση και τις υψηλές τιμές των αγαθών και των πρώτων υλών. Παραμένει υψηλή η τιμή του πετρελαίου, όπως γνωρίζετε, και αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση ε, στην οικονομική ανάκαμψη. Συζητήθηκε αυτό το θέμα και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ σήμερα το πρωί. Και εκφράσαμε όλοι τις ανησυχίες μας ακριβώς για αυτό το γεγονός, για τις τιμές του πετρελαίου που είναι ψηλά και συνεχίζουν να αυξάνονται. Επίσης, χρηματαγορές. Έχουμε ε, προβλήματα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα αναχρηματοδότησης κάποιων πιο αδυνάτων οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι τώρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι το θέμα μας σήμερα και θα πρέπει να το συζητήσουμε σε βάθος. Όπως γνωρίζετε όλοι, βασικό στόχος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να δοθεί μια ε, εκ των προτέρων σαφής διάσταση στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έρχεται να συμπληρώσει το ευρωπαϊκό επίπεδο τις Εθνικέ προσπάθειες για τους προπολογισμού με κατευθυντήριες γραμμές για πολιτικές πριν οι χώρε λάβουν οριστικές αποφάσεις για τον προπολογισμό του επομένου έτους. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα ευθυγραμμίσει στο Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη της πολιτικές παρακολούθησης εποπτείας και θα συντονίσει το χρονοδιάγραμμα. Ενώ νομικά ε, τα δύο αυτά θέματα δεν συνδέονται, είναι ξεχωριστά θέματα. Μακροοικονομική σταθερότητα, δημοσιονομική πειθαρχία και προσπάθειες που κάνουν τα κράτη ε, να ε, ευθυγραμμιστούν με τη στρατηγική του 2020. Η ετήσια έκθεση ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε, ε, δημοσιεύτηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2011 και έθεσε ε, σε τροχιά ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο που απαιτεί εκ των προτέρων και το τονίζω αυτό συντονισμό ε, τη οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών πριν όλα αυτά γίνουν δεσμεύσει στα κράτη-μέλη για τους προπολογισμού του 2012. Δέκα είναι οι δράσει που περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2011 και το 2012. Του προπολογισμού αντίστοιχα. Πάντα όλα αυτά εγγράφονται στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020. Στο Συμβούλιο έχουμε ήδη εγκρίνει το Φεβρουάριο συμπεράσματα για μακροοικονομικές πτυχές και δημοσιονομικές βάσει ε, της στρατηγικής για την ετήσια ανάπτυξη. Το Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, εντοπίσει τις ε, κοινέ προκλήσεις και θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Καλώς ορίσατε κύριε Ρεν, αγαπητέ, όλοι. Το είδα και το πρωί βέβαια, όλη η ώρα. Είναι πάντα μαζί μας όλοι και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, οι προσανατολισμοί αυτοί θα ληφθούν υπόψη όταν θα προετοιμάζονται τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης και τα εθνικά προγράμματα. Όλα αυτά μέχρι τον Απρίλιο. Τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα εθνικά σχέδια ε, μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σύγκλησης και σταθερότητας πάλι τον Απρίλιο. Θα τα αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο και τον Ιούνιο. Θα ε, προκύψουν κάποιες συστάσεις πολιτικής, αν αυτό χρειαστεί. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να τα πραγματοποιήσει όλα αυτά εγκαίρω, έτσι ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο να εγκρίνει γνώμε, νομοδοτήσει και συστάσεις αναχώρα. Θα πρέπει να λαμβάνουν αυτά πλέον τώρα τα κράτη-μέλη υπόψη, προετοιμάζοντα, καταρτίζοντα του προπολογισμού του για το 2012 και να τα συμπεριλαμβάνουν στις ε, ε, ιδέες και στο σχεδιασμό τους. Όπως γνωρίζετε, Θέλουμε όλα αυτά να αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να βεβαιωνόμαστε ότι de facto έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και για την οικονομία στα κράτη-μέλη. Τι θα συμβεί τώρα, δηλαδή σε μερικούς μήνες. Θα έχουμε μια ενσωματωμένη, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την οικονομική πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη μακροοικονομική σταθερότητα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών, πράγμα που είναι εκ των όνων κάνευ για να έχουμε μια ανάπτυξη βιώσιμη, ευφυή και που να συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι ένα εξαιρετικό μέσο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για μας, έτσι ώστε ταυτόχρονα να αξιολογούμε, να εκτιμούμε ε, κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι πολιτικές και ενισχύεται η ανάπτυξη και η δημοσιονομική κατάσταση όλων των κρατών μελών. Θα ήθελα να πω κάτι εμπαρόδο, σύντομα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναφέρω. Ήδη αναφερθήκαμε στις προοπτικές της οικονομικής μεγέθυνσης ή ανάπτυξης. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα ανεργίας, υψηλή ανεργία μεταξύ των νέων και αυτό δεν είναι βιώσιμο να φτάνουν δείκτες ανεργίες ε, το 20 και παραπάνω, 20 με 40% ανεργία των νέων σε ορισμένα Ιδιαίτερα τους νέους επαναλαμβάνω πλήττει ανεργία και θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης τονώνοντας ε, την ανάπτυξη της οικονομίας. Και τέλος, αν σας καταλαβαίνω καλά κυρία Πρόεδρε που μου κάνετε νοήματα, ε, θα ήθελα να πω ότι τα εθνικά μας κοινοβούλια και πολλοί από εσά σήμερα εδώ εκπροσωπείτε τα εθνικά μας κοινοβούλια ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στις πολιτικές που εκτελούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών πολιτικών και ως δημοσιονομική αρχή τα κοινοβούλια αποφασίζουν και ψηφίζουν τον προπολογισμό για τους πόρους που χρησιμοποιούν τα κράτη. Είμαστε λοιπόν στα χέρια των εθνικών μας κοινοβουλίων και ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είμαστε στα δικά σας χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι μας αρέσει να είναι οι υπουργοί στα χέρια του Κοινοβουλίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Ζαν Κλοντ Juncker που είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, κυρίες βουλευτές. Δεν ξέρω αν υπήρξαν πριν από μάνα πολλοί ομιλητές. Δεν αγνοείται πλέον τίποτα όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο για το τι ακριβώς θα γίνει οπότε δεν θα καθίσω τώρα να σας εξηγήσω λεπτομερώς για το περί τίνος πρόκειται. Εγώ συχνά είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με ευρωβουλευτές και με εθνικούς βουλευτές. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Οι παρόντες εδώ το ξέρουν όλοι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς κάνουμε. Εγώ θα κοιτάξω να είμαι σύντομος να πω απλώς ότι το θέμα και το περιεχόμενο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με ικανοποιεί, διότι από τότε είμαι πρόεδρος του Eurogroup δεν κάνω τίποτα άλλο από το να ε, υπερασπίζομαι να κάνω αγώνα για ένα τέτοιο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον αυτά τα οικονομικά να έχουμε σωστό διάλογο σε θέματα που αφορούν τους προπολογισμού και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν στις χώρες μέλη, ούτω ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις πολιτικές μας, τι δικέ μα και των αλλωνών, ούτω ώστε να γίνουν σεβαστά κάποια κριτήρια. Τώρα, σε σχέση με αυτό που υπήρξε, υπάρχει κάτι το καινούριο. Είναι το σύμφωνο του ευρώ. Αυτό εδώ, στην ουσία, είναι η επιστέγαση όλης της διαδικασίας διαβούλευσης και του συντονισμού που ξέρουμε μέχρι τώρα. Το σύμφωνο αυτό του ευρώ το οποίο θέλαμε στην αρχή να πούμε σύμφωνο για, την, για τον ανταγωνισμό, ανταγωνιστικότητα, ε, να εξασφαλίσουμε όλα τα μέσα τα οποία χρειάζονται ώστε να ενισχυθεί ο συντονισμός των οικονομικών μας πολιτικών. Ε, πρέπει, πρέπει, έχει γίνει κατανοητό ότι για να περάσουμε σε αυτό το σύμφωνο του ευρώ θα πρέπει να εισαχθεί όλη αυτή η στρατηγική στα πλαίσια του 2020 και με ενορχιστρωμένες κατευθυντήριες γραμμές όπου θα έχουμε όλες τις αρχές που έχουν ε, υιοθετηθεί όσον αφορά στο σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, όσον αφορά το θέματα του μέσου, έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε για να προχωρήσουμε καλύτερα. Να προσθέσω τώρα ότι το κείμενο που προτείνει η, ε, Επιτροπή τέλη του ε, Σεπτέμβρη 2010 έχει όλες τις ε, οδηγίες και όλα τα κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα, λοιπόν, από εδώ μέχρι τον Ιούνιο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, δείξει τη φιλοδοξία του για τα θέματα που αφορούν τη την οικονομική διακυβέρνηση και αν κατορθώσουμε μέχρι τέλη της επόμενης εβδομάδας να έχουμε ένα μηχανισμό σταθερότητας στην Ευρώπη. Αν πετύχουμε λοιπόν να διευκολύνουμε την ε, δημοσιονομική σταθερότητα και εδώ έχουμε και το θέμα της Ιρλανδίας είναι κατανοητό είναι μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτική και ποσοτική ε, συνέχεια και ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν με όλη αυτή τη διαδικασία επιτέλους ένα συνεκτικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε και κάτι το οποίο θα λέγαμε τόσο μα τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Τώρα για το σύμφωνο του ευρώ θα ήθελα να πω οι κυβερνήσεις επιτέλους καταλάβαν ότι δεν είναι πλέον τώρα, δεν έχουμε να κάνουμε, ε, να κάνουμε ποιηματάκια αλλά και να κάνουμε διάφορους καταλόγους Αντιθέτως, χρειάζεται μια αξιολόγηση ε, για να δούμε τι ακριβώς έγινε ή δεν έγινε στις διάφορες χώρες. Γι' αυτό το λόγο, ανάμεσα στους στόχους που έχουν ε, καθοριστεί με το σύμφωνο του ευρώ, οι, ε, οι πρωθυπουργοί, λέει το κείμενο, θα πρέπει να επιλέξουν κάποιες προτεραιότητες εθνικές. Η κάθε χώρα θα πρέπει να το κάνει αυτό μέχρι το ε, Μάρτιο, ούτως ώστε μέχρι τον Ιούνιο θα να έχουμε όλες τις, ε, την ενημέρωση, να ενημερωθεί η Κομισιόν για ποιες ακριβώς είναι οι προτεραιότητες. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε, να διασαφηνίσουμε όλες τις πολιτικές. Είναι γεγονός όμως ότι αυτό το σύμφωνο για το ευρώ δεν είναι. Έχει να κάνει με την αρχική ιδέα που είχε αναφέρει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκόζη, διότι κάποια στοιχεία έχουν εξαφανιστεί, έχουν... δεν υπάρχουν. Υπάρχουν διάφοροι στόχοι. Υπάρχει το θέμα των κυρώσεων και των εθνικών ε, αρμοδιοτήτων και των κυβερνήσεων στις χώρες μέλη. Θα δούμε λοιπόν όταν γίνει η αυτοψία, ε, γι' αυτό εδώ το για την εκροψία είπε ο πρόεδρος. Θα δούμε δηλαδή πώς έχει ακριβώ η κατάσταση, αν μπορεί δηλαδή να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ένα συντονισμό των ε, της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Ενδιαφέρονται τόσο οι ευρωβουλευτές όσο και οι εθνικοί βουλευτές. Θα υπάρχει μια συνάντηση 11 Μαρτίου και έχει γίνει μια πρόοδο, θα λέγαμε, ένα βήμα μπροστά, διότι αποφασίσαμε οι χώρε μέλη σε κάθε στάδιο ε, όταν θα υπάρχει η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα πρέπει ε, να βλέπουμε εκεί πέρα ότι θα γίνεται μια σωστή ε, συνέχεια και τήρηση των συστάσεων της Κομισιόν. Η δεμοί θα έχουμε και ένα σύστημα, αυτόματο σύστημα κυρώσεων. κάτι το οποίο υποστηρίξαν πολύ οι τρεις κυβερνήσεις των χωρών Μπενολούξ, διότι ο μόνοι τους και κυρίως ο πρόεδρος του Eurogroup έχει μια μεγάλη έννοια, ε, θέλει πραγματικά να υπάρξει μία πρόεδρος πρόοδος ε, να προχωρήσουμε, Αυτά σε γενικές γράμμες, κυρία Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα με ευχαρίστηση να ε, συζητήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Είμαι βεβαία ότι όλοι θα σκεφτούμε διάφορες ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις να σας υποβάλουμε. Τέλος, ε, περνάμε στον Επίτροπο για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα, τον κύριο Όλη Ευχαριστώ, Σάρον. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας πω ότι με μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτήν την επίκαιρη διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Sharon Bowles και την Επιτροπή ΕΚΟΝ και τα μέλη της, γιατί ανέλαβαν αυτήν την επίκαιρη πρωτοβουλία. Τόσο ο Γιώργη Ματόλσεν όσο και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σας έδωσαν τις απόψεις τους για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και για την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση και το σύμφωνο για το ευρώ. Οπότε θα είμαι σύντομος να συμπληρώσω μόνο κάποια πράγματα γιατί περάσαμε ένα, δύο μέρες όχι δύο μέρες και δύο νύχτες όπως συνήθως δύο μέρες στην ομάδα Eurogroup και συνδυάσαμε τις ευρωπαϊκές απόψεις όσον αφορά την οικονομική μας ανταπόκριση στην τελευταία φάση της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης να πω δύο λόγια για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ε, τι σημαίνει αυτό. Αλλά καταρχήν να πω κάτι για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης γενικότερα και για το ιστορικό στο οποίο βασιστήκαμε για να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία έδειξαν πως είναι και η ώρα να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση αν και τα πρώτα δέκα χρόνια του ευρώ ήταν επιτυχή. Εν γέννη, ωστόσο, η νομισματική η χρηματοπιστωτική κρίση τόνεσε κάποια προβλήματα στο σύστημά μας. και συνέβαλε μαζί με σφάλματα πολιτικής κάποιων χωρών στο να αυξηθεί η οικονομική αστάθεια στην Ευρώπη και να κινδυνεύει η οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε την κρίση που αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και σε κάποιες άλλες χώρες. Στην Ελλάδα βασικά πρόκειται για μια κρίση στην Ιρλανδία για τραπεζική κρίση και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα που έπαιξαν το ρόλο τους. Συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι χρειάζεται να βρούμε τέτοιου είδους μέσα ώστε να μπορούμε να εμποδίσουμε μια τέτοια κρίση στο μέλλον και να ενισχύσουμε το πολιτικό πλαίσιο στην οικονομική και νομισματική πολιτική της Ευρώπης. Τώρα, Τώρα, για το σύμφωνο περιλαμβάνει έξι νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ε, συνολική μας προσέγγιση στην κρίση, καθώς ενισχύει τόσο την προληπτική όσο και τη διορθωτική πτυχή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επεκτείνοντας το πεδίο της οικονομικής εποπτείας καθώς και την διόρθωση των μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών μέσω της βελτίωσης των μηχανισμών επιβολής και ενισχύοντας τα εθνικά μας ε, πλαίσια οικονομίας. Καθώς και προσδίδοντας στην Ευρώπη τα κατάλληλα μέσα που χρειάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπόρεσε το Συμβούλιο να συμφωνήσει για μια γενική προσέγγιση για το νομοθετικό πακέτο που θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μας με το Ευρωκοινοβούλιο ώστε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική εργασία μέχρι το καλοκαίρι. με όσο γίνεται πιο φιλόδοξη, έκβαση στις εργασίες αυτές. Και θέλω να ευχαριστήσω την Εγκρική Προεδρία για την εξαιρετικά επικοδομητική και παραγωγική εργασία της στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Πρέπει να πω ότι όταν η Κομισιόν ε, υπέβαλε τις ιδέες της και τις πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης την περασμένη άνοιξη, πριν από ένα χρόνο, επικράτησε σκεπτικισμός και δυστημία. Αλλά σήμερα, όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη εν γέννη στηρίζουν το πυρήνα των έξι νομοθετικών προτάσεων. Γι' αυτό και μιλάμε για ιστορική μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, που είναι στην καρδιά της οικονομικής διακυβέρνησης και που αρχικά προτάθηκε πριν από κάποια χρόνια από τον ε, πρωθυπουργο Ζαν Jean-Claude Juncker του Λουξεμβούργου, που κάθεται δίπλα μου, ε, και τον οποίο συγχαίρω για αυτήν την ε, φαϊνή ιδέα που είχε τότε. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία λοιπόν που, που τώρα έχει μετατραπεί σε πραγματικότητα και που θα είναι πολύ σημαντική για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Και αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση σε σχέση με το εξάμεινο. Η Κομισιόν εξ αρχής έχει τονίσει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν στην δημοσιονομική εποπτεία και προτείναμε να χορηγηθεί στην Κομισιόν και ενδεχομένως στο Συμβούλιο Αρμοδιότητες για την εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών παλιότερα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε ή ότι θα μπορούσαμε να εμπλακούμε στις λεπτομέρειες ε, και στις αποφάσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αντιθέτως, αυτό θα σημαίνει ανάλυση και παρακολούθηση από τους εταίρους των βασικών δημοσιονομικών ε, κατευθυντηρίων γραμμών, καθώς και εναρμόνιση της οικονομικής πολιτικής και των εθνικών προϋπολογισμών σε, σε δράση συντονισμού η, ανάλυση, η Κομισιόν θα αναλύει πριν από την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών και θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε συστάσεις και να αναμένει διορθωτικές ενέργειες. Ορισμένοι επέκριναν αυτή την πρόταση, ότι δηλαδή πρόκειται για παραβίαση της κοινοβουλευτικής κυριαρχίας. Εγώ ίδιος είμαι πρώην μέλος ενός εθνικού ε, Κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ευαισθησίες ε, των ε, δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων των κοινοβουλίων. Δεν θέλουμε να παραβιάσουμε τη δημοκρατία καθόλου. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα σεβαστούν τους ίδιους κανόνες που τα ίδια αποφάσισαν στην συνθήκη και στο σύμφωνο. Δηλαδή στην ουσία να κάνουν αυτό που διακηρύσουν ότι θα κάνουν. Και σε σχέση με τις επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όσον αφορά τις μελλοντικές εργασίες, είναι ένα στοιχείο της συνολικής οικονομικής στρατηγικής που αποτελείται από την ε, οικονομική παγίωση, την ανάπτυξη της μεγέθυνσης, διευθυντικές μεταρρυθμίσεις καθώς και ολοκλήρωση την, ε, της οικονομικής μας κατάσταση. Όπως είπε και ο Γιάννη Κλόντ Γιούνκερ, την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο αναμένεται να λάβει αποφάσεις κλειδιά για αυτή την πολιτική και να δώσει και πολιτικές κατευθύνσεις για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, μελλοντική εργασία στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και της εποπτείας αυτής. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω συνοψίζοντας τα εξή ότι οι η διακυβέρνηση μάλλον και οι μετα... πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει αποκομίσει τα σωστά διδάγματα από την κρίση και ενεργεί πλέον σύμφωνα με αυτά με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ωστόσο, ένα επιτυχές αποτέλεσμα, δηλαδή το ξεπέρασμα της κρίσης δεν είναι εγγυημένο και είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε την ελαφρώς βελτιωμένη μακροοικονομική εικόνα να μας οδηγήσουν σε υπερβολές, υπέρματρες φιλοδοξίες. Αν ενεργήσουμε σοφά και αποφασιστικά σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να αντιστρέψουμε την τάση να, ξεπεράσουμε το σκόπελο και ε, αν το περσινή χρονιά ήταν ε, χρονιά κρίσης και επιβίωσης, η φετινή χρονιά μπορεί να αποτελέσει τη χρονιά της μεταρρύθμισης και της αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Um, I have... Και εγώ σας ευχαριστώ και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει το λόγο μόλις δύο συνάδελφοι. Θέλει και... Ωραία, τρίτος και μέλη και της Επιτροπής ε, Οικονομικών και Νοσμικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α, τώρα καταφθάνουν όλοι γρήγορα, γρήγορα. Από τη γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας πρώτα, ο κύριος Σεφτσικ, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα ομαδοποιήσουμε μερικές ερωτήσεις και μετά θα επανέλθουμε για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεται να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέματα που είναι κυρίως διακυβερνητικά. Και, ε, εκτιμώ ε, αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε εμείς οι βουλευτές μεταξύ μας. Ωστόσο, πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά μέτρα που θα λάβει μετά από 10 μέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εμείς δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Σε τι συνίστανται. Δεν θα μπορούσε ο κύριος Ρεν ή ε, άλλοι προσκεκλημένοι να μας διευκρινίσουν λίγο περισσότερο περί τίνος πρόκειται, τι θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι μέτρα θα εγκρίνει. Εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν Πρωθυπουργό που στις, την 11η βραδινή θα έχει μπροστά του μια απόφαση να λάβει πριν τα μεσάνυχτα ή πριν τις 2 το πρωί για θέματα τόσο ουσιαστικά, τόσο κομβικά, με τέτοια πίεση χρόνου. Από τον Ιανουάριο είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε την κρίση έτσι. Λέμε ότι λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα για να ληφθεί η επόμενη κρίση. Η σημερινή όμως κρίση, τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται περιμένουμε να λυθεί από μόνη της. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ και καιρό, να μην σας πω καθημερινά, θα μπορούσατε να μα δώσετε λοιπόν πιο συγκεκριμένε λεπτομέρειε τι μέτρα επίκειται να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά από 10 μέρε. Για να ξέρουμε ότι η λογοδοσία θα παραμένει στα πολιτικά όργανα, εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί ακούμε μεγάλα λόγια πριν τις εκλογές και μετά ερχόμαστε απέναντι σε ελλείμματα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Από τη Λιθουανία, ο κύριος Ανδρεκάτης. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ήθελα να επιμείνω σε μια σειρά πτυχών του θέματος. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για μέτρα τα οποία καλύπτονται ήδη από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του, της Συνθήκης της και, άλλα και άλλων κειμένων. Δηλαδή μιλάμε για επικάλυψη εδώ πέρα. Θα πρέπει να το δούμε. Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία δηλαδή. Οι χώρες του ευρώ και οι χώρες που είναι εκτός βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις οι χώρες που είναι εκτός της Ευρωζώνης έχουν διαφορετικά νομίσματα, έχουν συστήματα και τράπεζες εντελώς διαφορετικά. Η Λιθουανία, για παράδειγμα, βρίσκεται σε μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τη Πολωνία. Το εθνικό νόμισμα στην Πολωνία φέρει π μπορεί να υποτιμηθεί. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε στη Λιθουανία. Ήτι, ε, μπορεί να κάνει να βγάλει το συμπέρασμα ότι εδώ έχουμε διαφορές ουσιώδεις. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο μήπως δυσκολεύει τα πράγματα για την ένταξη στο ευρώ για κάποιες χώρες. Μας ανησυχεί. Απ' την άλλη υπάρχουν και άλλα θέματα που τίθενται. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το κοφίν. το θέμα του ελέγχου για τον προπολογισμό είναι σημαντικό. Αλλά το, ε, ο έλεγχο εξ είναι εξίσου σημαντικός για μας. Είναι σημαντικό για τα εθνικά κοινοβούλια για να ξέρουμε πώς μπορούμε στα εθνικά κοινοβούλια να έχουμε όχι μόνο ε, και τους δύο δυνατού ελέγχους. Υπάρχει θέμα ευθύνη. Αυτό θα μπορέσει να μας επιτρέψει να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε όσον αφορά τον σεβασμό, τη δέσμευσή μας απέναντι σε πράγματα για τα οποία όντως έχουμε δεσμευτεί. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος ε, ε, σημείωσε αυτά που ρωτάτε και για το Σύμφωνο Σταθερότητας και λέτε ότι υπάρχει μια επικάλυψη με άλλα θέματα. Ίσως χρειάζεται να επανέλθουμε για κάποιες απαντήσεις ε, σε αυτές τις πρώτες ερωτήσεις. Χρόνο έχουμε, δεν χρειάζεται να συλλέξουμε όλες τις ερωτήσεις. Όλοι, θέλεις να απαντήσεις για το σύμφωνο. Thank you. Actually, Ευχαριστώ. Εγώ ε, σου έκανα νοήματα γιατί δεν έβλεπα τον ομιλητή και ήθελα να μου πεις που κάθεται. Ε, δεν ήταν για να απαντήσω. Σε αυτό το θέμα νομίζω είναι πιο ενδεδειγμένος να απαντήσει ο Ζαν Κλοντ Ιούγκερ ως ε, πρόεδρος του Eurogroup. Διότι αυτό αποφασίστηκε Σύνοδο Κορυφής τη Ευρωζώνης και εκείνο ήταν εκεί και έπαιρνε τι αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, όντω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις σε όλα τα μέτωπα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση για την εξυγίανση των προϋπολογισμών Βέβαια αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά να δεσμευτούν ε, να ανταποκριθούν στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για παράδειγμα η Πορτογαλία έχει λάβει πάρα πολύ ουσιαστικά μέτρα και αποφάσεις για την εξυγίανση του προπολογισμού και διαρθρωτικά μέτρα τις ε, προηγούμενες ημέρες, καθώς επίσης και κάποιες άλλες χώρες. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική συμφωνία για ε, την ίδρυση του μονίμου πλέον μηχανισμού ε, σταθεροποίησης που θα αντικαταστήσει τον προσωρινό. Και επίσης ε, τη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση και να ολοκληρωθούν και οι δοκιμές αντοχής των τραπεζών, αυτά τα stress test και αν χρειάζεται να αναδιαρθρωθεί το θέμα της ε, ε, αύξησης κεφαλαίου των τραπεζών και των πιστοτικών ιδρυμάτων. Για να αντιμετωπίσουμε, δεν θα έλεγα τα τελευταία στάδια της κρίσης, τα πιο πρόσφατα στάδια της κρίσης. Η κρίση αυτή γνωρίζετε ότι από τη φύση της είναι κρίση χρέους σε κάποια κράτη-μέλη ε, ε, σε κάποια άλλα μέρη της Ένωσης παραμένει σοβαρή τραπεζική κρίση. Εσείς οι βουλευτές όταν μελετάτε την ευρωπαϊκή οικονομία και τις οικονομίες των κρατών μελών διαπιστώνετε ότι πραγματικά, η πραγματική οικονομία ε, ανασυντάσσεται και γίνεται και πιο ανεξάρτητη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσεται και απασχόληση, η οποία δεν είναι ακόμα βέβαια. Έχουμε κάποιες αναταραχές στις χρηματαγορές και πρέπει να τις συγκρατήσουμε. Αυτά θα αποφασίσει την άλλη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ. Έρθουμε τώρα στο Jean-Claude Juncker. Μήπως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε και για το πώς πηγαίνει η πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί συμφωνία της Παρασκευής αργά το βράδυ, του Σαββάτου το πρωί. Ίσως οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας θέλουν να το διαμορφώσουμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες αυτό που σε γενικές γραμμές αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Μάλιστα, για να απαντήσω στον συνάδελφο από τη Λιθανία. Ναι, και εγώ το διατύπωσα με τον ίδιο τρόπο. Το σύμφωνο για το ευρώ ή για τον ανταγωνισμό όπως ανταγωνιστικότητα όπως είπατε δεν προσθέτει κάποια δεν έχουμε κάποια προσθέμενη αξία πάνω σε αυτό. Η δική μου εμπειρία είναι τέτοια ε, πολλές φορές ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει σαν ένα κύμα να διαχυθεί χωρίς χωρίς να καταλάβει κανείς γιατί προκαλούνται όλα αυτά τα διαδοχικά κύματα. Διότι έχουμε το Σύμφωνο ανάπτυξης και τις μεγάλες μεγάλε οικονομικού προσανατολισμού, κατευθυντήριε γραμμέ που διαμορφώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την απασχόληση. Εμείς εξετάζουμε σε κάθε συνεδρία του Eurogroup την κατάσταση κάθε χώρας μέλους κάνουμε συστάσεις αναχώρα των χωρών μελών της Ευρωζώνης για να επανορθώσουν επανορθώσει ενδεχομένως την πολιτική τους. Αναρωτιέται κανείς αυτό το σύμβολο τώρα για το ευρώ τι, για ποιο λόγο γίνεται. Υπάρχουν ε, κάποιες εξηγήσεις που θα μπορούσα να σας δώσω. Ο λόγος είναι χρειάζεται να μαζέψουμε σε μια ενιαία διαδικασία όλα τα διαφορετικά, τα επιμέρους θέματα και ιδέα. Γιατί αυτή είναι η ιδέα της Συμφώνης της Ευρώς. Να ανατεθεί το θέμα της διακυβέρνησης από, δηλαδή να ανατεθεί αυτό το θέμα της διακυβέρνησης από τους ίδιους τους αρχηγούς κρατών και μελών και σε θέματα που έχουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις είναι μια νέα, ξέρετε, ιδέα διότι παλιά οι, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας είχαν τους ελέγχους και όλα τα ανάλογα. Να σας πω τώρα ποια είναι η δική μου επιθεση. Δεν είναι σαφές, δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει. Δεν είναι δεδομένο, σας το λέω ειλικρινά. Ας φανταστεί κανείς. Οι 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντιούνται με τους υπόλοιπους και να συζητήσουν λεπτομερώς όλες οι ιδιαιτερότητες προ, προβλήματα που αφορούν, από τα, αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια και να συνδυάσει κανείς και να δει τις λύσεις των μεν και τις λύσεις που προβλέπουν οι άλλοι, να γίνουν συγκρίσεις, τους ρυθμούς, το ένα, μεταρρυθμίσεις, το άλλο, όλα αυτά τα θέματα κατάρτισης, θέματα μισολογικά, μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ενδεχομένως πρέπει να γίνουν, ειλικρινά αυτή η διαδικασία μας ξεπερνάει. Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί κάτι. Φερρυπίν. Η κυρία Μέρκελ, έτσι λένε, εγώ δεν το είδα ποτέ, δεν είδα κάποιο έγγραφο επίσημο γαλλογερμανικό, δεν ξέρω δηλαδή ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Φαίνεται λοιπόν, λέγεται, ότι η Γερμανία θα πρότεινε να καταργηθεί το σύστημα φορολόγησης που υπάρχει στο Λουξεμβούργο και στο, Βούλιο, και στο βελιό. και όταν, όταν είδα αυτή την ιδέα και τη συζήτησα με κάποιους συναδέλφους είπα για πείτε μου ποια είναι η διαφορά ανάμεσα τις, ανάμεσα στις διαφορές που έχουμε ανάμεσα στο σύστημα το βελικό και το λουξεμβουργιανό. Δεν είχαν ιδέα. Δεν ξέραν καν ότι υπάρχουν διαφορέ. διαφορές. Δεν τους επικρίνω διότι κάποιοι υπουργοί δεν ξέρανε ότι στις χώρες τους Φερρυπίνη σε θέματα ε, μηχανισμών ε, ε, συλλογικών συμβάσεων δεν ξέρανε ακριβώς πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα. Πώς θα διαπραγματευτούν δηλαδή. Τη στιγμή που δεν ξέρει καθόλου για το δικό του σύστημα πώς θα λειτουργήσει ο άνθρωπος αυτός να, να, επι, να κριτικάρει, να έχει απόψη για κάποιο άλλο σύστημα. Λοιπόν, είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο δεν θα μπορέσει να οδηγήσει πουθενά. Δηλαδή μου προκαλεί αλλεργία ε, να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορεί να έχει κάποιος που να τα ξέρει όλα. Τον Ιούνιο 2005 σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Είχαμε, ξέρετε ότι είχαμε συζητήσει για ένα σύμφωνο, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νεότητα. Εγώ το ξέρω το. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Θεωρήθηκε ίσως ότι ήταν το πιο πολύ σημαντικό θέμα. Το... Είχε γίνει πολύ μεγάλο με την πανοκρουσίαση, είχε λασαριστεί αυτό το σύμφωνο για την νεότητα. Κανείς δεν το θυμάται. Αν επιμένουν δηλαδή οι πρωθυπουργοί να θέλουν να επιμένουν σε κάτι ανάλογο για το ευρώ, πραγματικά δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Η Επιτροπή, η Κομισιόν θα πρέπει να παίξει το ρόλο της και τα διάφορα όργανα του Συμβουλίου, το ΕΚΟΦΗΝ, το Eurogroup πρέπει να έχουν το δικό τους ρόλο. Είναι υποχρεωμένοι κατά με. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία να δει κανείς πώς μπορεί κανείς να, διαφε... να προκαλέσει ενδιαφέρον των εθνικών κοινοβουλίων για αυτό το σύμφωνο. Υπάρχει μία ε, ε, διευκρίνηση όσον αφορά τις μεθόδους, υπάρχουν κάποιοι στόχοι που έχουν προταθεί από το σύμφωνο για το ευρώ και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα θέμα που αφορά την Ευρωζώνη. Είμαι πεπισμένος ότι οι χώρες μέλη που έχουν το ίδιο νόμισμα έχουν ανάγκη από ένα συντονισμό. Αλλά να πω επίσης να μην δημιουργήσουμε ένα καινούριο χάσμα χώρες ευρώ από τη μία, κυβερνήσεις των μεν, κυβερνήσεις των χωρών που είναι εκτός. Όχι ένα καινούριο τείχος ανάμεσα στις χώρες που έχουν το υιοθετήσει το ευρώ και από τις άλλες που είναι εκτός. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οι φίλοι μας από τη Λιθουανία, την Πολωνία και άλλοι έχουν απαιτήσει οι 15, οι 17 της Ευρωζώνης να μην δουλέψουν μόνοι τους για την, συντονισμό της ε, κοινή ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Το κάναμε αυτό και για το, μηχανισμό της, ε, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τη Σταθερότητα. Τέλος πάντων, το σύμφωνο για το ευρώ θα πρέπει να μην είναι τέτοιο το οποίο θα οδηγήσει σε μια, μια ένα αντίθεση ανάμεσα στις χώρες που είναι στην Ευρωζώνη και σε άλλες που είναι εκτό, εκτός. Η, η ζώνη ευρώ δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ. Όλες οι χώρες που εκπληρώνουν τα κριτήρια θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. Όλες, επαναλαμβάνω, ε, οι εγώ πιστεύω ότι οι χώρε οι οποίε εκπληρώνουν τα κριτήρια θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να ενταχθούν στο ευρώ. Όχι δηλαδή αν το θέλουν ή όχι, υποχρεωτικά θα πρέπει να περνάνε στο ευρώ. Ξέρω ότι οι βουλευτέ από τη Σουηδία έχουν μια άλλη άποψη. Έχουμε να κάνουμε εδώ και με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Υπάρχουν κάποιοι όροι εκεί ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επιβάλλει και έναν έλεγχο και φυσικά εδώ το θέμα του ελέγχου ex post είναι αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων Δεδομένου όμως ότι τόσο στα, Ευρωπαϊκά, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο, στην Ευρώπη θα πρέπει να συζητήσουμε για τις ε, μεταρρυθμίσεις που ενδεχομένω να χρειάζονται. Τίποτα άλλο όσον αφορά την προστιθέμενη αξία. Thank Well, uh, and... Σας ευχαριστώ πολύ. ξέχασα κάτι. Ρωτήσατε για τη συνέχεια που θα δοθεί, που δόθηκε μετά από το Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής. Εχθές ε, συγκέντρωσα την, ε, το Eurogroup για να συζητήσουμε τα θέματα που έμεναν ανοιχτά θα πρέπει να δούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ευρώ, δηλαδή οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των 17, έχουν προοδεύσει γιατί αποφασίσαμε να αυξήσουμε την πραγματική δυνατότητα δανεισμού της στα 440 δις και προβλέψαμε να φροντίσουμε στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουνίου 2013 να ανέλθει στα 500 δις αλλά σε επίπεδο Συμβουλίου του Ευρώ, δηλαδή σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, δεν είχαμε συζητήσει διάφορες λεπτομέρειες εκτός από το pricing για την Ελλάδα, όπου συμφωνήσαμε για την Ελλάδα ότι έπρεπε να μειωθεί το επιτόκιο για την Ελλάδα. με βάση την διάρκεια απόσβεσης, αποπληρωμής, συγγνώμη, από πλευρά των ε, ελληνικών αρχών που ήταν 7,5 χρόνια. Αλλά δεν είχαμε μιλήσει ούτε για την ε, διευκόλυνση, ούτε για το μηχανισμό, ε, δεν είχαμε μιλήσει για τα μελλοντικά επιτόκια, για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δεν είχαμε συζητήσει για τους κανόνες διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και θα πρέπει να πω ότι σε επίπεδο Eurogroup δεν προχωρήσαμε πολύ γιατί κυρίως για τη δομή του κεφαλαίου του Μηχανισμού Σταθερότητας οι απόψεις των κρατών μελών είναι αρκετά αποκλίνουσες πράγμα που με έκανε να συγκαλέσω εκ νέου το Eurogroup για την επόμενη Δευτέρα είναι μια συνεδρίαση όπου θα συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη. Κανονικά ο Ούγκρος Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να προεδρεύσει αυτή τη ομάδα, αλλά εφόσον πρόκειται για παράνομη συνεδρίαση, γιατί είναι μια συνεδρίαση όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια συνεδρίαση των εκπροσώπων των 27 κρατών μελών, γιατί συζητάμε στην Ευρώπη για έναν διακυβερνητικό μηχανισμό που είναι εκτός συνθήκων, οι συνάδελφοι δεν βρήκαν τίποτα καλύτερο να κάνουν παρά να τον αλλάξουν αυτόν που ήθελε να έχει ένα τέτοιο μηχανισμό και να μας οδηγήσουν να, να, να, να αναθέσουν μάλλον σε κάποιον άλλον να φτιάξει αυτόν τον διακυβερνητικό μηχανισμό. Τη Δευτέρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε για τα εκκρεμή ζητήματα, ώστε το Συμβούλιο 24 και 25 Μαρτίου να μπορέσει να κλείσει το θέμα Νομίζω πως είναι απολύτως απαραίτητο να ε, διατυπωθεί μια άντιση στην κρίση του χρέους στη ζώνη του ευρώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και θα πρέπει αυτό να γίνει με τρόπο που να μην είναι κάτω από τον, ο, τις προσδοκίες των αγορών. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα στο επίπεδο της Ευρωζώνης είναι ότι είμαστε πάντα πίσω σε σχέση με τις απόψεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αν ήμασταν πιο ευέλικτοι, πιο έτοιμοι, πιο γρήγοροι, πιο εφευρετικοί και φάνταστοι, θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί των αγορών. Όσο είμαστε πίσω, τιμωρούμεθα. Την ημέρα που θα μπορέσουμε να προηγηθούμε, τότε θα τιμωρηθούν οι ε, αγορές. Περιμένετε λοιπόν τη ρεβάνση. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, διαβάζετε τις δικές μου ομιλίες και απαντάτε με βάση αυτά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουν κι άλλοι. Πρώτα, τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη σειρά που ζητήσατε το λόγο. Ο κύριος Χουντής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι οι συγητές, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που έκαναν, μου δημιούργησαν περισσότερες συγχύσεις και περισσότερες ανησυχίες για όλα αυτά που βλέπουμε ότι γίνονται μπροστά μας. Είχα την ευκαιρία να ξαναπώ ότι η σύγχυση στο επίπεδο των πολιτών είναι μεγάλη. Οικονομική διακυβέρνηση, ευρωπαϊκό εξάμεινο, σύμφωνα ανταγωνιστικότητας, σύμφωνο που δεν το λέμε ανταγωνιστικά και το λέμε σύμφωνο για το ευρώ και αναρωτιέται κανείς. Πρώτο, όλα αυτά που συζητούνται είναι μήπως εκτός των άλλων επί της μεθόδου μια μάχη εξουσίας, μια μάχη ισχύω μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπής Συμβουλίου με χαμένους και θύματα αυτής της διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια των οποίων η γνώμη δεν ζητείται. Ερώτηση πιο συγκεκριμένη πείτε ότι σε ένα εθνικό κοινοβούλιο απορρίπτεται το σύμφωνο για το ευρώ. Τι θα προκύψει. Ερώτηση δεύτερη. Το σύμφωνο για το ευρώ μήπως εμπεριέχει μια έμεση τροποποίηση των συνθήκων γιατί μπαίνει σε χωράφια που δεν περιλαμβάνονται στις συνθήκες και τότε υπάρχει θέμα νομιμότητας και συμβατότητας με τις συνθήκες. Οι ερωτήσεις αυτές θα μπορούσαν να καταλήξουν, εν πάση περιπτώσει, τελειώνω με μια ερώτηση είναι φανερό ότι όλους με αυτούς τους συντονισμούς και τις πειθαρχίε, επιτρέψτε μου το σχόλιο, ένα συντονισμό, ένα σύμφωνο για να λυθεί το πρόβλημα της αυξανόμενης ανεργίας για την Ευρώπη δεν βλέπουμε. Αυτό θα προκύψει. Πείτε ότι όλος αυτός ο συντονισμός γερμανικής έμπνευσης καταφέρει να γίνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης, της Ευρωζώνης και κατά, μικρές Γερμανίες. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο όραμα. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να δώσει λύση στα προβλήματα που έχει συνολικά η Ευρώπη. Σταματώ εδώ γιατί θα σας κουράσω με τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Thank you very much. And next... Ευχαριστώ. Από την Αυστρία τώρα ο κύριος Στούμπολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ που έχουμε αυτό το σύμφωνο για το ευρώ τώρα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη εκπλήρωση του. Βεβαίω. η πολιτική ξέρουμε ότι είναι η τέχνη του εφικτού και πολλές φορές το εφικτό είναι ο ελάχιστος κοινό παρονομαστής. Έχουμε μάθει από τον τύπο τις προθέσεις Μέρκελ και Σαρκοζή και για λόγους ρεάλ αυτά ήταν καταδικασμένα να αποτύχουν. Εγώ διαπιστώνω ότι έχουμε σε πολλά κράτη-μέλη πρόβλημα επικοινωνίας, ε, εντυνόμενο συνεχώς με τους πολίτες μας που στο κάτω-κάτω είναι και ψηφοφόροι μας. Εγώ πώς θα βγω να εξηγήσω. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Είναι αρκετά δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν έχουμε κρίση του ευρώ αλλά κρίση ορισμένων κρατών του ευρώ. Γιατί κάθε μέρα διαβάζουν για μηχανισμό διάσωση του ευρώ. Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι κοιτάξτε, το ευρώ είναι ισχυρό νόμισμα. Τα προβλήματα τα έχουν μερικέ χώρε μόνο. Και τώρα έχετε το επιχείρημα και μα λέει. Μα εξηγήσει τα κριτήρια του Μαστρίχ, το σύμφωνο σταθερότητα, στρατηγική τη Λισαβόνα. Όλα αυτά μα είπατε ότι θα πετύχουν. Και τώρα έρχεστε και μα λέτε το σύμφωνο για το ευρώ θα πετύχει. Και ρωτώ, εγώ τώρα τι να βγω να πω στον κόσμο, στου ψηφοφόρου μου για ποιο λόγο είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό που φτιάξαμε τώρα είναι πιο επιτυχές από όλα αυτά που είχαμε φτιάξει προηγουμένως. Εκτός από το να σας πω ότι για μια ελπίδα ζούμε. Ευχαριστώ. Άλλος ένας ακόμα και μετά απαντήσεις πάλι. Από την Ελλάδα, η κυρία Παπανδρέου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητέ. και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφόρων θεσμικών οργάνων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Ε, σίγουρα τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στο γίγνεσθε της Ευρώπης γιατί δεν πολύ ενδιαφέρονται και πρέπει να πω ότι η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, όλα αυτά είναι έννοιες πολύ μακριά για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Ε, και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και μπορεί εσείς να παίρνετε κάποιες αποφάσεις ε, που πιθανόν να αυξάνουν την γραφειοκρατία ή να αυξάνουν την σταθερότητα στην Ευρώπη αλλά αυξάνει αυτόχρονα και η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, είπατε ότι είστε πολύ ευχαριστημένος κύριε Γιούγκερ γιατί έχει ένα, ε, δημιουργήθηκε ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ε, διακυβέρνηση. Ε, θέλω σίγουρα ο συντονισμός είναι απαραίτητος. Έχω όμως την εντύπωση ότι η Ευρώπη, και αυτό δεν είναι δική μου εντύπωση, είναι γενικότερα, η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις too little, too late. Και κάθε φορά οι αποφάσεις που, παίρνουν, που παίρνονται δεν έχουν την επίδραση που θα ανέμενε κανείς. Προχθές το Συμβούλιο Κορφής πήρε κάποιες αποφάσεις. Ε, δεν ξέρω αν αυτές, κατά τη γνώμη μου, δεν λύνουν το πρόβλημα της Ευρώπης και δεν μιλάω για το πρόβλημα της Ελλάδος που είναι γνωστό, το πρόβλημα της Ευρώπης και σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να ξαναπάρουμε ή να ξαναπάρετε πάλι καινούριε αποφάσεις. Δεν δημιουργείται, δεν δίνεται μία οριστική λύση στο πρόβλημα του ευρώ, στο πρόβλημα της ε, Ευρώπης. Ε, σίγουρα η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη. Σίγουρα η εποπτεία είναι απαραίτητη. Μα αρκεί όμως αυτό. Το μόνο το πρόβλημα της Ευρώπης είναι απλώς δημοσιονομικό και σε έναν βαθμό έγινε δημοσιονομικό γιατί στήριξε αφιδωλώς και έτσι έπρεπε το τραπεζικό σύστημα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ε, είδαμε ότι το 2010 τα head funds είχαν <clears throat> πρωτοφανή κέρδη. Τα bonus και τα τοξικά ξανακυκλοφορούν. Η Ευρώπη δεν βλέπω να έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα και δεν γίνεται μόνο η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες για να εποπτεύσει, να βάλει κανόνες, αγοράς, κανόνες σε αυτή την, ε, την αγορά. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν το κόστος και κάποιοι βεβαίως κερδίζουν από την, ε, από την κρίση. Για την ανάπτυξη μας λέτε τώρα πάλι είναι η προοπτική του Growth Stability Pact για το 2020. Έγινε κάποια ανάλυση γιατί η Λισαβόνα δεν ε, πέτυχε. Και τι μας διασφαλίζει ότι θα πετύχουμε τώρα. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπιστεί την Κίνα, την Ινδία. Υπάρχει το πρόβλημα της Ιαπωνίας τώρα, υπάρχει ο αραβικός κόσμος που είναι σε αναστάτωση. Αυτά τα πράγματα τα έχει κανείς ε, μελετήσει και δει το τι συνέπειες και το τι πρέπει να κάνουμε. Ε, με ποιο τρόπο, αν απλώς ο στόχος μας είναι να μειώνουμε το χρέος και τα ελλείμματα, θα γίνουμε κάποτε, όπως λέγόταν πρωτοπόροι σε θέματα έρευνας και καινοτομίας ε, έχουμε υποχρέωση να πληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά όχι μόνο χαμηλότερα ελλείμματα και χαμηλότερο χρέος, αλλά να τους κληρονομήσουμε και υποδομές και συστήματα υγείας και συστήματα εκπαίδευσης. Και με τις περικοπές που βάζουμε συνεχώς, δεν ξέρω εάν το χρέος μας προς τις επόμενες γενιές μειώνεται ή μεγαλώνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση από την Άστρικ Λούλινγκ από το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Γιούνκερ που τόσο καλά έδωσε το σχετικό χαρακτήρα αυτού του συμφώνου για την Ευρώπη. Γιατί εγώ Αφελώς ε, σκέφτηκα ότι αυτό το six pack, τις έξι προτάσεις της Κομισιόν όπως αποκαλέστηκε την ενίσχυση της ε, οικονομικής ε, πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής είναι, είναι σπάνιο. Επ' αυτής της πρότασης θα έπρεπε να εστιάσουμε την προσοχή μας και να Ε, οδηγηθούμε σε συνένεση ώστε να υιοθετηθούν ε, από, με τη διαδικασία συναπόφασης γιατί όπως σας είπα αφελώς ε, πίστεψα ότι αυτά θα έπρεπε να βρίσκονται στην καρδιά των δικών μας, του δικού μας προβληματισμού και του προβληματισμού του Συμβουλίου. Τώρα μας έρχεται αυτό το περίφημο σύμφωνο για το ευρώ και δεν ξέρω πια με τι, τι να πιστέψω γιατί βρίσκω ότι κατ' ουσίαν αυτό που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και να μας απασχολήσει είναι οι προτάσεις της Κομισιόν και να φτάσουμε σε μια ε, γερή, δυνατή συμφωνία και θέλουμε να συμβάλλουμε εμείς εδώ το Κοινοβούλιο για μια τέτοια πρόταση. Φυσικά, συνεχίζουμε να τα συζητάμε όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να πω πως, ε, πώς να το πω τώρα έτσι κάπως διπλωματικά, είναι κάπως δύσκολο ε, είμαι κάπως έκπληκτη σε σχέση με αυτή τη στροφή που παίρνουν τα πράγματα. Να πω όμως, και σήμερα το πρωί είχαμε τη μεγάλη χαρά να συναντήσουμε την κυρία Λαγκάρντα και τον κύριο Σόιμπλε. Και ο κύριος Σόιμπλε μας είπε ήδη πόσο μεγάλες προσπάθειες θα κάνει η Γερμανία. Μίλησε για κάτι δις για να χρηματοδοτηθεί ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Τώρα, αλήθεια, το μερίδιο που θα δοθεί σε κεφάλαια σε αυτό το σύμφωνο, αν κατάλαβα πολύ καλά τα πράγματα δεν είναι ακόμα και τόσο ξεκάθαρα, είναι δισεκατομμύρια που οι χώρες θα πρέπει αμέσως να εκταμιεύσουν. Θα ήθελα να το ξέρω. Γιατί εγώ είπα, ναι εντάξει μην κάνετε έτσι, δεν χρειάζεται να τα εκταμιεύσετε και αμέσω. Δεν ήταν πολύ ικανοποιημένος από τη δική μου ε, παρέμβαση και με ρώτησε αν ήμουν και εγώ εχθές στο ΕΚΟΦΗΝ. Μήπως λοιπόν μπορείτε εσείς να μας διευκρινίσετε πώς, τι, ποιο θα είναι το βάρος για κάθε χώρα όσον αφορά την συνεισφορά τους ε, με κεφάλαια σε αυτόν τον μηχανισμό σταθερότητας. Ε, επίσης, Ακούσαμε διάφορα κοπλιμέντα από την κυρία Λαγκάρντ σε σχέση με την θέση του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά την φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ξέρετε πως μια πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υιοθέτησε μια τέτοια πρόταση, αλλά δεν έγινε λόγος μόνο για την Ευρωζώνη. Όμως σήμερα το πρωί η κυρία Λαγκάρντ μας είπε ότι πιστεύει πως αυτό ο φόρος θα πρέπει να ισχύσει μόνο για την Ευρωζώνη. Δεν ξέρω πόσα δώρα θέλετε να κάνετε ακόμα στον κύριο Κάμερον, αλλά θα μου το πείτε. Τώρα, για τα ευρωομόλογα, εντάξει, γίνεται ντόρο για αυτά. Οι Γερμανοί όταν τα ακούν δεν θέλω αλλά θα σα πω εγώ ότι η συζήτηση για τα ευρωομόλογα ε, έχει πάρει μέγεθο ε, ε, πολέμου, θρησκευτικού πολέμου πια. Αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πια υιοθετώντα το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση και δεν πιστεύω πως είναι λογικό να προβλεφθεί αυτό το μέσο απλά και μόνο για να χρηματοδοτηθεί το χρέος με καλύτερα επιτόκια, πράγμα που θέλουν να εξασφαλίσουν διάφοροι, ενώ ταυτόχρονα όλοι γνωρίζουμε ότι σε κάποια φάση η προσφυγή στα ευρωομόλογα μπορεί να είναι υποχρεωτική. Εσείς ε, ή ο κύριος Ρέν μπορείτε να μας πείτε ή να ορίσετε ποιες θα είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η προσφυγή σε ευρωομόλογα να αποτελέσει κάτι το φυσιολογικό και ποιο θα είναι το απαραίτητο ποιοτικό άλμα που θα πρέπει να γίνει προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, Καλό είναι να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις. Ε, δεν νομίζω πως όλοι πρέπει να απαντήσουν σε όλα. Ελπίζω πως όταν θα έχετε ολοκληρώσει ε, και οι τρεις σας θα έχετε δώσει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Σάρων. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το εξή. Συμφωνώ απολύτως. 100% με τον Αυστριακό συνάδελφο ότι δεν πρόκειται για κρίση του ευρώ είναι η χρηματοοικονομική κρίση ε, ορισμένων οικονομιών, ορισμένων κρατών της Ευρωζώνης. Σε κάποιο βαθμό, αυτό ήθελα να πω και εγώ, τα προβλήματά μας προέρχονται από την τεράστια επιτυχία του ευρώ, διότι απεδείχθη τεράστια επιτυχία του ευρώ τα τελευταία 12 χρόνια τώρα. Ας κοιτάξουμε στο παρελθόν τι γινότανε. Το 99 ήρθε το ευρώ και προχώρησε δυναμικά, ενισχυόταν όλο και περισσότερο και μετά μια ωραία ημέρα δέχτηκε επίθεση από την ε, παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Δεν είμαστε εμεί οι ένοχοι. Ο πραγματικό ένοχο είναι η τεράστια επιτυχία του ευρώ. Είναι θύμα τη επιτυχία του το ευρώ. Και αυτό σε τι οφείλεται. Δεν υπάρχει κάτι που να ορίζεται ως ομοιογενής ευρωπαϊκή οικονομία. Και το χρηματοοικονομικό ε, σύστημα δεν είναι ενιαίο παντού στο παρασκήνιο πίσω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό το λόγο εμείς οι Ευρωπαίοι, οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι, οι υπουργοί προσπαθούμε να χαράξουμε μία συνολική απάντηση ε, σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των συνθήκων, και αυτό είναι ένα τμήμα της ολοκληρωμένης απάντησης, αν θέλετε. Το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση, τα έξι νομοθετήματα, προσπαθούν και αυτό να είναι ένα τμήμα της συνολικής ολοκληρωμένης απάντησης για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, που είναι το θέμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή ή ένα από τα θέματα, το ευρωπαϊκό εξάμεινο και όλη η διαδικασία για πιο ισχυρή και πιο επιτυχή ε, οικονομική πολιτική και καλύτερο συντονισμό είναι και αυτό τμήμα, ένα τμήμα της συνολικής απάντησης. Το σύμφωνο για το ευρώ και το σύμφωνο για τη σταθερότητα. Και πάλι είναι ένα τμήμα και μόνο του ενιαίου εγχειρήματο που καλύπτει ολόκληρη την οικονομική διακυβέρνηση και τη συνολική απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Ο κανονισμός για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η σχετική διαδικασία και αυτό είναι ένα στοιχείο. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Σάρων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πραγματικός ένοχος των προβλημάτων που γνωρίζουμε σήμερα είναι η τεράστια επιτυχία του ευρώ την τελευταία 12 ετία. Και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να πετύχουμε. Με μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που να υποστηρίζει όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Είμαστε στο μετέχνιο δηλαδή. Προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε μεγαλύτερο βαθμό ε, συντονίζεται η οικονομική πολιτική, αλλά σταδιακά και βήμα-βήμα. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια ακόμα, μερικά χρόνια για να επιτύχουμε και να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη πλέον και ενοποιημένη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ελπίσουμε όμως το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές από τις ερωτήσεις απευθύνθηκα άμεσα ε, σε σένα, Ζαν Κλόντ, αν θέλεις να απαντήσεις. Να απαντήσω πρώτα στις ερωτήσεις. για να ε, που θα αφήσω για τον Όλη να απαντήσει. Δηλαδή θα μοιραστούμε μεταξύ μας τις διάφορες ερωτήσεις, τα διάφορα θέματα, ποιος θα απαντήσει σε τι. Λοιπόν, Όλοι, νομίζω πρέπει να απαντήσεις για τον κανονισμό. Γιατί είπε η Βάσο ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά στη ρύθμιση του κανονισμού και επειδή έχει εν μέρη δίκιο θα προτιμούσα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα, θα ήθελα να πω στον κύριο Χουντή, στον Έλληνα συνάδελφο εκεί, η άκρα αριστερά, ότι το σύμφωνο για το ευρώ είναι σύμφωνο που έχει συναυθεί μεταξύ κυβερνήσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Συνδέει τις κυβερνήσεις μεταξύ τους αυτό το σύμφωνο ε, των χωρών της Ευρωζώνης και ενδεχομένως εκείνων που κάποια στιγμή θελήσουν να ενταχθούν. Οι κυβερνήσεις που συνήψαν αυτό το σύμφωνο υπόκεινται σε ένα εθνικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν ξέρω πώς ε, γίνονται αυτά αλλού, αλλά στη δική μου χώρα γίνονται ως εξής. Πριν έρθουμε στο Συμβούλιο των 17, πριν έρθω εγώ προσωπικά, με κάλεσε το κοινοβούλιο μου στην Ολομέλεια και χρειάστηκε να εξηγήσω ποια θέση θα υπερασπιζόμουν στις Βρυξέλλες για το σύμφωνο για το ευρώ. Επειδή η θέση σε ισχύ του συμφώνου για το ευρώ υποχρεωτικά περνάει μέσα από τα εθνικά συστήματα μεταρρυθμίσεων, την επομένη κάλεσαν τον Υπουργό Οικονομίας στο Κοινοβούλιο ακριβώς για να εξηγήσει τα στοιχεία και τους στόχους που θα έβαζε στο Εθνικό Πρόγραμμα για τις Μεταρρυθμίσεις. Τον Απρίλιο, όταν συνεδριάσει ε, τέλη Μαρτίου το Συμβούλιο, θα ε, έχουμε και άλλη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής μας, όπου θα κληθεί η κυβέρνηση να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της ή για τις παραλήψεις της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και όπου διαφωνεί η Βουλή του Λουξεμβούργου στα όσα έκανε η κυβέρνηση δεν θα απορρίψουν το σύμφωνο ε, για το ευρώ, αλλά μπορεί να ρίξουν την κυβέρνηση. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Είναι υπόλογε οι κυβερνήσει στη Βουλή του, στο εκάστοτε κοινοβούλιο. Και το κοινοβούλιο αποφασίζει αν έχει την εμπιστοσύνη η κυβέρνηση ή όχι. Και η λογική συνέχεια είναι το σύμφωνο του ευρώ, για το οποίο σα είπα πολλά καλά αλλά και πολλά κακά, αλλά δεν χρειάζεται περαιτέρω αναθεώρηση της συνθήκης. Η συνθήκη αναθεωρήθηκε για να μπορέσουμε να θέσουμε σε ισχύ το μηχανισμό, αυτό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και Σταθεροποίησης, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη μεταρρύθμιση και αναθεώρηση της συνθήκης, διότι ό,τι έχει να κάνει με το σύμφωνο για το ευρώ, ήταν και στην ατζέντα της Λισαβόνας ήδη, αλλά ε, είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη των κρατών. Συντονιζόμαστε, συμφωνούμε για κοινού στόχους και μετά θα ε, υιοθετήσουμε τα εθνικά μέτρα που θέλει ο καθένας να επιβάλλει στη χώρα του και να εφαρμόσει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που αναφέρονται λοιπόν σε αυτό το σύμφωνο για το ευρώ, τα οποία όλα στο σύνολό τους ήδη περιλαμβάνονται σε μια δήλωση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 1997 για την ενίσχυση της οικονομικής πολιτικής. Δίνουμε τώρα μια νέα μέθοδο στην οικονομική διακυβέρνηση. Διαπιστώσαμε ότι η ατζέντα της Λισαβόνας, θυμηθείτε, γιατί είμαστε στο 2011 και αν θυμάστε μέχρι το 2010 έπρεπε να είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι ή πιο ανταγωνιστική ε, ήπειρος του κόσμου. Εγκρίναμε την ατζέντα της Λισαβόνας με την Πανοκρουσίες. Αλλά θυμάστε το τραγούδι «Παρόλε, παρόλε, παρόλε». Γιατί οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν υπό το κράτος της ε, ατζέντα της Λισαβόνας δεν έγιναν. Έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις μένα, αλλά όχι όλες όσες έπρεπε να γίνουν. Γιατί δεν έγινε καμία αξιολόγηση. Δεν υπήρχε όργανο που να ερχόταν να παρακολουθεί, να κοιτάει τι γίνεται με τη Λισαβόνα, πώς προχωρεί. Το σύμφωνο λοιπόν για το ευρώ είναι, αν θέλετε, ένα εγχειρίδιο μεθόδου για να εργάζονται οι ε, πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις για να ελέγχουν πώς εφαρμόζονται αυτά τα ε, μέτρα. Δεν πρόκειται να γίνει από μόνο του. Σε σχέση με το παρελθόν, πρώτα απ' όλα, είναι νέα η μέθοδος αυτή. Οι κυβερνήσεις αλληλοεπιτηρούνται και με πολύ πιο αυστηρό βλέμμα από ό,τι στο παρελθόν. αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να πω ότι δεν θα γίνουμε όλοι μικρές Γερμανίες. Εγώ έχω άλλες πατριωτικές φιλοδοξίες από αυτή. Εξάλλου, ένα μεγάλο δουκάτο δεν μπορεί να γίνει μια μικρή Γερμανία. Δεν θα υποβαθμιστούμε κιόλα για να σας κάνουμε τη χάρη. Είμαστε, εμείς είμαστε μεγάλο δουκάτο, δεν θα γίνουμε μικρή Γερμανία και να ε, ε, κοπούμε σε περιφέρειες. Χαίρομαι ήδη πάρα πολύ που έχουμε λιγότερες περιφερειακές εκλογές στο Μεγάλο Δουκάτο από τη Γερμανία. Γιατί είναι πιο εύκολο να κυβερνάει κανείς χωρίς ε, αυτό το αέναο ε, περιφερειακό γίγνεσθε και τις εκλογές και τις επιρροές. Έχουμε 12 επαρχίες, 12 καντόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε κάθε τρεις και λίγο νέα κυβέρνηση σε κάθε καντόνι. Γιατί θα ήταν λίγο έτσι αταξία και παραφωνία αυτό. Λοιπόν, έχουμε τους ίδιους στόχους και με τους Γερμανούς και με τους υπολείπους, αλλά δεν είμαστε ε, ε υπό καμία εντολή ούτε γερμανική, ούτε γαλλική, ούτε βρετανική, ούτε τίποτα, δεν ξέρω. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε και ξέρετε τι έχουμε ξεχάσει στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μάθουμε ξανά την τέχνη και την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση να θέλουμε να συνεργαζόμαστε γιατί μαζί πρέπει να προχωρήσουμε. Ακούω τις συζητήσεις και στο Eurogroup και αλλού. Η λέξη Ευρώπη δεν εμφανίζεται ε, αρκετά συχνά. Όλοι εξηγούν και εγώ έτσι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους αλλά επειδή είμαι πρόεδρος απλώς προεδρεύω και το κλείνω και αφήνω τους άλλους να μιλάνε. Λοιπόν, όλοι έρχονται και εξηγούν γιατί δεν μπορεί να το κουνήσει κανείς πιθαμή, γιατί με βάση την εθνική του άποψη και τα λοιπά έχουμε το αβ πρόβλημα, το γ, το δ. Και ερχόμαστε να θρήσουμε όλα τα εθνικά προβλήματα και ποτέ δεν βρίσκουμε λύση, ευρωπαϊκή όμως. Θα πρέπει να ξαναμάθουμε να αγαπάμε ένα τον άλλον. Ε, το έχουμε ξεχάσει αυτό θα πρέπει να θέλουμε περισσότερη Ευρώπη για να υπάρξει μια στοιχειώδης, μια ελάχιστη. Αν θέλουμε όλη ελάχιστη Ευρώπη θα εύχομαι περισσότερα έθνη κράτη. Ε, αυτό είναι ε, στην ουσία αυτό που ισχύει η πραγματικότητα. Όλοι, θα απαντήσεις στην κυρία Λούλινγκ σε παρακαλώ για τα 500 δισεκατομμύρια ή μια που έχω ξεκινήσει τώρα να τα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, μιλώ υπό τον έλεγχο του Όλη Ρεν θα πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο πρώτα, το πώς, για να φτάσουμε σε μια δυνατότητα ε, δάνεια εδώ της 500 δις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να συλλεγεί αυτό το κεφάλαιο. Το Συμβούλιο των 17 είπε, και δεν ήταν κανένα έβριμα αυτό, ότι θα πρέπει να είναι ένα τμήμα ε, κεφαλαίο, ένα τμήμα έχει εγγύησεις και ένα τμήμα callable. Μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο callable και το guarantees, τις εγγύησεις. Το callable δεν ξέρω τι διαφορά έχει από τις εγγύησεις. Θα δούμε πώς θα μεταφερθεί αυτό στην πράξη. Ε, σας επισημαίνω δε ότι θέλουμε να δώσουμε πραγματική δυνατότητα δανειοδότησης στο μηχανισμό. Θα πρέπει να είναι ε, τα 500 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Τη Δευτέρα θα το συζητήσουμε για το πότε και πώς. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση κεφαλαίου, αν μου επιτρέπετε, της διευκόλυνσης ε, του σταθεροποιητικού μηχανισμού. Διότι εκεί είχαμε προβλέψει 440 δις, αλλά δεδομένης της κατάστασης και των εγγύσεων που έπρεπε να δώσουμε, πρέπει να πέσουμε σε ένα άλλο πόσο, φτάσαμε στα 250 περίπου δις και πρέπει να ξαναφτάσουμε στα 440. Και σίγουρα αυτό θα γίνει μέσω εγγύησεων. Παρόλο που μερικοί θεωρούν ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα που να πληρώνουν οι χώρες που δεν είναι τριπλό α. Και πάλι όλα αυτά είναι υπό έλεγχο, υπό εξέταση. Φαίνεται ότι συζητήσατε με τον κύριο Σόιμπλε και σας το έχω ξαναπεί στο παρελθόν κυρία Λούλινγκ. Όταν χάνετε τον προσανατολισμό σας στη ζωή, να ε, κοιτάτε τον Πρωθυπουργό σας που έχει μεγάλα ατού και μπορεί να σας ε, διασκεδάσει κάθε φόβο και κάθε αγωνία που μπορεί να έχετε. Τα ποσά λοιπόν που θα στείλουμε στο μηχανισμό σταθεροποίησης μετά από απόφαση που πρέπει να λάβει Eurostat, που είναι ανεξάρτητη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να δει αν αυτό εντάσσεται στο δημόσιο χρέο ή όχι των κρατών μελών. Αν αυτό ο μηχανισμός σταθεροποίηση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός, ανεξάρτητος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που θα τον συναπαρτίζουν τα κράτη-μέλη και θα έχει μια δομή διακυβέρνηση, που θα αποδεικνύει όμως ότι έχει αρκετά μεγάλη αυτονομία, τότε οι κεφαλαιακές ε, ενέσεις αυτές δεν θα θεωρηθούν ε, τμήμα του χρέους, αλλά επένδυση, αν θέλετε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Αλλά στο εσωτερικό δίκαιο ε, δημοσιονομικού του προπολογισμού στη Γερμανία, στο εσωτερικό της Γερμανίας το συνυπολογίζουν ως τμήμα του ελλείμματος. Ακόμα και αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν το μετράνε στο χρέος, στη Γερμανία το προσμετρούν στο ε, ε, έλλειμμα, το ετήσιο έλλειμμα, το ταμιακό με βάση την αμυγή λογιστική. Αυτό έπρεπε να σας είχε απαντήσει ο κύριος Σόιμπλε που δεν σας τα είπε. Όλοι για την στρατηγική για το 2010 θα μας πεις κάτι, έχεις να μας πεις κάτι. Ναι. Νομίζω πως ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ διαλέγει τις καλύτερες ερωτήσεις, πιο εύκολες και αφήνει τα ζώρικα για μένα. Αλλά είμαι ευγνώμων που ο πρόεδρος του Eurogroup μου δίνει το λόγο τελικά. Μπορώ κι εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις ακόμα, μα θέλεις. Ε, πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά εδώ πρέπει να βρούμε λύσεις. Καταρχήν για την ερώτηση της κυρίας Λούλινγκ για τα ευρωομόλογα. <laughs> Καταλαβαίνω γιατί ο Ζαν Κλόντ μου ρίξε τον μπαλάκι γι' αυτό το θέμα. Θα πρέπει να πω ότι ανέκαθεν θεωρούσα ότι τα Eurobond ήταν μια πνευματικώς ε, ελκυστική ιδέα. Είναι κάτι πολύ ευρύ που καλύπτει πολλές δυνατότητες όσον αφορά εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης των ε, δυνητικών ευρωομολόγων. Πρόσφατη πρόταση του, της ομάδας προβληματισμού Μπρούγκελ που μοιράζει τα ομόλογα σε μπλε, κόκκινα, πράσινα που μπορεί δηλαδή να καλύψουν ε, χρηματοδότηση που θα είναι κάτω από το επίπεδο των κριτήριων της Μάστριχ του 60% του ΑΕΠ ε, θα ήταν ένα είδος μπλε ευρωμολόγων αυτά, ενώ όταν ξεπεράσει αυτά βρίσκεσαι μόνος σου και πληρώνεις πιο, πιο ψηλά επιτόκια. Τα κόκκινα ομόλογα είναι αυτά, που είναι εθνικά ομόλογα, σύμφωνα με αυτή την ε, λογική. Όμως δεν λειτουργούμε εν κενό, αντιθέτως ε, βρισκόμαστε σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση κρίσης και γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις. Μπορώ να σας πω ότι κάναμε μια πρόταση τον Μάιο πέρυσι, σε 9 Μαΐου μάλιστα, το Σαββατοκύριακο μετά από το ελληνικό πακέτο και κατά τη διάρκεια εκείνης της εβδομάδας οι αγορές Είχαν ε, περάσει μεγάλη αναταραχή, τα σπρέτ ήταν πολύ μεγάλα, τα επιτόκια είχαν εκτοξευθεί και το Ευρωγκρούπ, Υπουργοί Οικονομικών και Κομισιόν αν είχαμε αναλάβει το έργο της ε, δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αυτό που κάναμε λοιπόν σε εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν να προετοιμάσουμε μια πρόταση. Βέβαια τη βγάλαμε από το σιρτάρι, προσαρμόσαμε, την προσαρμόσαμε και κάναμε μια πρόταση για έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας επί τη βάση δύο στοιχείων. Πρώτον, με εγγύηση του προπολογισμού της Ένωσης, ως ένα κοινοτικό δηλαδή μέσο, το πρώτο τμήμα μέχρι το κατόφλι των 60 δις του προϋπολογισμού δηλαδή της Ένωσης, επί τη βάση της εγγύησης του προϋπολογισμού της Ένωσης δηλαδή και μετά επί τη βάση κοινή εγγύησης από διάφορα κράτη-μέρη. Όλα αυτά μέσα στο πολύ κομψό πλαίσιο της ε, λήψης αποφάσεων ε, της κοινότητας. Το πρώτο κομμάτι υιοθετήθηκε και αποτελεί σήμερα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ενώ το δεύτερο τμήμα αναθεωρήθηκε εκ βάθρων και μετετράπη σε μια διακυβερνητική ε, ρύθμιση που είναι η διευκόλυνση ο μηχανισμός μάλλον ο ευρωπαϊκός για την ε, οικονομική διευκόλυνση. Γιατί λοιπόν δεν μιλήσαμε για ευρωομόλογα, γιατί ακριβώς αυτά έπρεπε να συνοδεύονται από διάφορες εγγύησεις και η πρόταση αυτή απορρίφθηκε. Και άρα στο τέλος αναγκαστήκαμε να δεχτούμε διακυβερνητική ρύθμιση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτήν τη ρύθμιση στιγμή που δημιουργήθηκε. Αυτό είναι το ιστορικό και άρα λοιπόν σε αυτή εδώ τη συγκυρία επειδή δεν βλέπω να είναι όριμες οι πολιτικές προϋποθέσεις για οποιοδήποτε ευρωμόλογο, οι προσπάθειές μας εστιάζονται στην δημιουργία του μόνιμου μηχανισμού για τη σταθερότητα που θα αρχίσει να ισχύει από τον Ιούνιο του 2013 και μέχρι τότε με την ενίσχυση της ε, δυνατότητας δανεισμού του FSF ώστε να έχουμε έναν τρόπο για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, μελλοντική κρίση. Τώρα, για τα διάφορα ταμεία τους διάφορους μηχανισμούς σταθερότητα, και τη ε, μέσο διευκόλυνσαν και δεν υπάρχουν εδώ συμπατριώτες μου, δεν υπάρχουν Φινλαδοί στην διάσκεψη εκεί, γιατί είναι απλό, γιατί έχουμε εκλογές σε λίγες εβδομάδες και δεύτερον, σε αυτή τη στιγμή η φιλανδική κυβέρνηση αυτή την ώρα μάλιστα έχει να αντιμετωπίσει μια πρόταση μορφής από την αντιπολίτευση λόγω της δημιουργίας του μηχανισμού και της επιβολής του EFSF. Άρα λοιπόν μη σας εκπλήσει που δεν υπάρχει κανείς εδώ από τη Φιλανδία. Είναι όλοι στο Κοινοβούλιο και συζητάνε γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα, την πρόταση μορφής. Για να συμπληρώσω τώρα τα όσα είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, να σας πω ότι κατά την άποψή μου πρέπει να ολοκληρώσουμε την εργασία μας για μια πολιτική συμφωνία μέχρι την επόμενη Πέμπτη Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γι' αυτό και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ συγκάλεσε την έκτακτη συνεδρία του Eurogroup την επόμενη Δευτέρα και είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί η πολιτική συμφωνία μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Μετά από την πολιτική συμφωνία στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Μαρτίου, η νομική συμφωνία για το ESM και για οι τροποποιήσεις για το EFSF, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν συμφωνηθεί 440 εκατομμύρια ως ε, πραγματική δανειστική δυνατότητα, θα ολοκληρωθεί ομαλά στις επόμενες εβδομάδες και η εθνική διαδικασία να ολοκληρωθεί και για τις δύο συμφωνίες ταυτόχρονα μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα σαφέ πρόγραμμα εργασία. Σα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ελπίζω να μπορείτε όλοι να το υποστηρίξετε, γιατί να θυμίσω ότι. Για να τα πω ειλικρινά, αυτό ήταν η άλλη όψη του συμφώνου και της συνολικής ανταπόκρισης που αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα από την διάσκεψη κορυφής της Ευρωζώνης και αναμένω να εγκριθεί και από το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Με άλλα λόγια, η μία πτυχή ήταν η εντατικοποιημένη οικονομική παγίωση, ιδιαίτερα από το Συμβούλιο αναμένεται να το κάνουν οι πιο ευάλωτες χώρες. Η Ισπανία το έκανε, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ε, για την ε, εξυγίανση και για τις διευθυντικές πολιτικές. Έχουν αναλάβει υποδεσμευτικά μέτρα. Δούλεψαν, δουλέψαμε πολύ στενά για τρεις εβδομάδε μαζί με τον Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλές άλλες χώρες ξεκίνησαν σε αυτή την ίδια πορεία εξυγίανσης και την επιτάχυνση των διαφορετικών αλλαγών, μεταρρυθμίσεων. Αυτό λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθεί από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά ε, χρειαζόμαστε ε, αρκετά σχηματική οικονομική σταθερότητα ώστε να δείξουμε ότι το short selling δεν είναι επικερδές σε σχέση με το ευρώ και γι' αυτό και οι φορείς της αγοράς λαμβάνουν υπόψη ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη και για να προστατεύσουμε την οικονομική ανάκαμψη και να βελτιώσουμε την απασχόληση στην Ευρώπη. Πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες μα. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνο να λες στους πολιτικούς ότι έχει σχεδόν εξαντληθεί η λίστα γιατί ξαναγέμισε αμέσως. Λοιπόν, θα ομαδοποιήσουμε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις και θα ακολουθήσουν σύντομες απαντήσεις. Θα σας πω ποιοι είναι στην ουρά. Αυστρία. Χριστόφ Μάξενέτα, Γερμανία. Βάιντινγκ και Μπράκμαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Ποδηματά, Ντομένιτσι, Καλχάιντ Λούντ, Γερουσαλόμ και Βίκυ Φόρτ. Και εσύ, Λίζα, και Λίζα Φερέρα. Άλλος, κανείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι. Μπορεί να κλείσει εδώ. Α, η κυρία Χιούβνερ. Καλώς. Να κλείσει ο κατάλογος, πρέπει να βιαστούμε τώρα. Πρώτα εθνικά κοινοβούλια, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους έχουμε συχνά ως θύματα εδώ τους ημερινούς εκπροσώπους. Εσείς δεν τους βλέπετε τόσο πολύ συχνά. Χρήστοφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τα ειλικρινή του σχόλια, λέει ο κύριος Ματσνέτερ. Δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση, αλλά και χρήματα αγορές βλέπουν ότι κάθε εβδομάδα Έχουμε μεγαλύτερε εξαγγελίε και νέε εξαγγελίε για νέα πακέτα, για νέους μηχανισμούς, για νέα διάσωση και αυτό προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση παρά λύνει τα προβλήματα. Και όπως είπε, σερνόμαστε πίσω από τις χρηματαγορές, έχουμε μείνει πίσω, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να κοιτάνε και τι αγορές κατάματα σε ίδιο επίπεδο. Τι είδαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Μια τραπεζική κρίση και δυστυχώς δεν έφταιγε η Ευρώπη. Τελικά πρότεινε ο Σαρκοζή, η Μέρκελ και ο Στάινμπρουκ ε, να δράσουν πυροσβεστικά και το καταφέρανε, ε, έδρασαν πυροσβεστικά και σώσαν τις τράπεζες. Ταυτόχρονα όμως ο συντονισμός των κρατών μελών δεν λειτουργήσε ε, αρκετά καλά αλλά στη συνέχεια ήρθαμε και σώσαμε ε, το 2009 τα πράγματα, ε, τουλάχιστον να περιορίσουμε ε, τη μείωση της πραγματικής οικονομίας και το στραγγαλισμό της οικονομίας. Καταφέραμε αυτό να το αποτρέψουμε. Ωραία. Και μετά έχουμε μια κατάσταση όπου η επιπλέον χρέωση τώρα των κρατών μελών που απορρέει από αυτή την κατάσταση έχει γίνει αντικείμενο μιας τεράστιας σπέκουλας και κερδοσκοπίας. Καλά, οι Έλληνες λένε ότι το ελληνικό κράτος είναι χρωμένο τα τελευταία 3.500 χρόνια, ε, αλλά ε, χρειάστηκε να δώσουμε ε, δισεκατομμύρια και, ε, και τρέχαμε να τα βρούμε και οι δικές μας ευρωπαϊκές τράπεζες συμμετείχαν στο παιχνίδι αυτό. Ή εκείνοι που κάναν τη μόχλευση για τα μεγάλα ταμεία και μέσω του CDS ε, οδηγούσαν στα τα επιτόκια για να βγάλουν δισεκατομμύρια. Βλέπουμε το αποτέλεσμα στους ισολογισμούς των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, hedge funds κτλ. Τι τεράστια κέρδη έχουν. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, όπου η ίδια πυροσβεστική γίνεται εμπριστής. Μας έχουν φέρει σε τέτοια κατάσταση χρέους, ακριβώς λόγω των αποφάσεων και πολιτικά αυτά είναι αφόρητα, διότι σε τελική ανάλυση όλοι, ε, δεν ξέρω αν είμαστε βουλευτές, κυβερνώντες, υπουργοί και διεθνώς δρόντες, όλοι είμαστε εκπρόσωποι ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Και είναι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και πληρώνουν τρεις φορές για το ίδιο πράγμα. Αυτή που είναι το last resort, η τελευταία λύση. Δεν μπορούμε να, κάνουμε περικοπές στα κοινωνικά, να αυξάνουμε τους φόρους, να σώνουμε τις τράπεζες και τελικά να πληρώνει τη διαφορά και πάλι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος για τρίτη φορά γιατί έχουμε επιτόκια 700, 800, 900 και CDS και spread. Ποια είναι η πολιτική ανάπτυξη Ποια είναι η πολιτική ε, απάντηση. Το είπε και ο Γιούγκερ. Η ε, Ευρώπη μπορεί να γίνει αυτό. Ας πούμε, ευρωμόλογα. Εγώ είμαι ένας ταπεινός οικονομικός ελεγκτής και έχω και μια μικρή πείρα. Α, όλοι γνωρίζουν ότι εάν πέντε άνθρωποι από κοινού εγγυώνται για ένα δάνειο, είναι χαμηλότερος ο κίνδυνος για τον δανειολήπτη παρά για τον καθένα από τους πέντε αυτούς που εγγυώνται το δάνειο. Αυτό το σημείο πρέπει να το δούμε και να το εξηγήσουμε και στους Γερμανούς φίλους, γιατί θα χρειαστούμε και μια τέτοια κοινοτική αλληλεγγύη. Αν συνεχιστεί η οικονομική κρίση που θα συνεχιστεί μετά τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία, ε, να δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη, από πού θα χρηματοδοτούμε τα μεγάλα έργα υποδομής. Γιατί για αυτά δεν πρόκειται να βρούμε τα χρήματα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που είναι τόσο υπερχρεωμένοι. Θα χρηματοδοτουμε τα μεγαλα εργα υποδομης γιατι γι αυτα δεν προκειται να βρουμε τα χρηματα απο τους εθνικους προυπολογισμους που ειναι τοσο υπερχρεωμενοι θα ηθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία που είχαμε να το συζητήσουμε σήμερα και παρακαλώ η συζήτηση που άρχισε σήμερα να συνεχιστεί και να ενταθεί και στο μέλλον, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε νέα ε, κοινοτικά ευρωπαϊκά μέσα. Ένα τελευταίο, ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, Πρόεδρε σερνόμαστε πίσω από την κερδοσκοπία των CDS. Και τελικά δεν μπορούμε ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ιρλανδία να ε, τρέχουμε να αγοράζουμε και να σώνουμε γερμανικές, γαλλικές, αυστριακές τράπεζες. Δεν έχουμε τα χρήματα ιστοδυνικές να το κάνουμε. Και ρωτάω και τον Όλη και τον Ζαν Κλοντ. Δεν μπορούμε να υπέβουμε στις αγορές για τα credit default swaps, να τους κόψουμε τα πόδια εκεί, να σταματήσουμε, να τα συζητήσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουν κεντρικές τράπεζες όταν υπάρχει κεντροσκοπία κατά του νομίσματός τους. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Τώρα είμαστε υπό χρονική πίεση, οπότε συντομεύετε αν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Ο κύριος Μπίντι. Θα προσπαθήσω. Δεν θέλω να μιλήσω για non-paper που δεν τα έχει διαβάσει κανένας και για τις συλλογικέ συμβάσεις στη Γερμανία είναι το τοπίο τόσο περίπλοκο ώστε κανένα συνάδελφο στο κοινοβούλιο να το έχει καταλάβει. Αυτά για τις παρατηρήσεις που κάνατε προηγουμένως για τις συλλογικέ συμβάσεις. Δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε αυτή η ηρωνία που είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι κυβερνώντες ή κάποιοι βουλευτές που δεν ξέρουν τι συμβαίνει στις συλλογικέ συμβάσεις της χώρας του. Εν πάση περιπτώσει. Έρχομαι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης και ε, τη χρηματοδότηση. Αναφερθήκατε σε τρεις πηγές. Είπατε το κεφάλαιο που καταβάλλεται, paid in capital. Το δεύτερο είναι εγγύησης και το άλλο, αυτό που είπατε τι ήτανε. Το callable. Ότι είναι κεφάλαιο που πρέπει να κινητοποιούνται. Πού θα βρεθούν αυτά, ρωτώ. Τι εννοείτε, ότι κάπου πρέπει να το βρούμε, όχι να το ψάξουμε, να το βρούμε. Πού θα το βρούμε το κεφάλαιο αυτό και ποια θα είναι η δομή, ποιος θα πληρώνει εκεί και οι αξιολογήσει πώ συνδέονται με αυτό και οι βαθμολογίε. Γιατί να σα εξηγήσω ένα αντανακλαστικό. Όταν ακούω τριπλό Α, σκέφτομαι αυτέ ε, του οίκου αξιολόγηση. Και μόλι ακούσω οίκο αξιολόγηση, χάνω την εμπιστοσύνη μου στο σύστημα. Γιατί αυτό που έμαθα είναι ότι αυτό που εκτιμούν αυτοί οι οίκοι είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Αλλιώ δεν θα είχαμε οδηγηθεί μέχρι εδώ. Ε, καλωσορίζω τις προτάσεις του κυρίου Ρεν, γιατί είναι προτάσεις νομοθετικές, είναι προτάσεις κοινοτικές και είναι προτάσεις εφαρμόσιμες. Μ' αρέσουν αυτά όλα. Και τέλος, θέλω να συμφωνήσω και με τον αυστριακό συνάδελφο. Θέλω λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα να μας πείτε. Αφηρημένα επί των αρχών συμφωνούμε όλα τα ηθικά, τα δεοντολογικά, τα σημειώνουμε. Η αγορά όμως δεν δίνει σημασία σε αυτά και συχνά θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι χώρες χειρίζονται φόρους, οι τράπεζες χειρίζονται καταθέσεις, οι ε, ασφαλιστικές εταιρείες χειρίζονται ε, εισφορές. Ε, όλοι με ξένα χρήματα και με διάφορους κινδύνους και ρίσκα. Και εμείς πολιτικοί ερχόμαστε και τα χειροκροτούμε. Τι ωραία, τι θαυμάσια. Χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Και όλα αυτά ε, που συμβαίνουν στην οικονομία γίνονται σε επικράτεια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με διαδικασίες που δεν θα ήταν επιτρεπτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να τα ρυθμίζουμε καλύτερα αυτά. Αφήστε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο θέμα του κράτους ή των τραπεζών. Στην Ελλάδα ήταν κρίση προϋπολογισμού. Για κοιτάξτε τι ρόλο έπαιξε στην Ελλάδα η Goldman και η Sachs. Εκεί να δείτε πώς συνδέεται το θέμα του τραπεζικού τομέα και η διαπλοκή της τράπεζας με το κράτος. Γιατί πρέπει ένα κράτος να, δέσει, να, να σώσει οπωσδήποτε μία τράπεζα. Οι ασφάλειες. Ε, βέβαια για γνωστούς και εύλογους λόγους η Ευρώπη δεν μπορούσε να αφήσει τις τράπεζες ε, χωρίς διάσωση. Αλλά βλέπουμε ότι την άλλη εβδομάδα συνεδριάζει και στην παρανομία μάλιστα ένα μικρό γκρουπ που δεν ε, είναι επίσημο όργανο για να αποφασίσει για αυτό το μηχανισμό διάσωσης. αυτό, αυτή την παράθεση για το παράνομο δεν το λέω εγώ, το παραθέτω, εσείς το είπατε. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί είναι ένα πράγμα που δεν μπορώ να εξηγήσω στον κόσμο, στους ψηφοφόρους. Όταν λέμε ότι μια χώρα είναι πολύ χρεωμένη και δεν προσμετράται αυτό στο ευρωπαϊκό χρέος. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου ότι δεν το προσμετράμε. Θα το εξήγησε και ο Σόιμπλε ήδη. Ο καθένας θα πει ότι βεβαίως στη Γερμανία αυτό θα είναι συν δύο δι. Ο κόσμος αισθάνεται ευθύνη για αυτό το πράγμα. Πώ θα του τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράχμαν από τη Γερμανία και πάλι. Παρακαλώ περιορίστε το χρόνο σας γιατί δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός Ματόλτσι προηγουμένως σωστά είπε ότι το ευρώ ευτυχώς ε, ε, είναι ένα νόμισμα επιτυχές και τίποτα άλλο. Βεβαίως είχε μεγάλη επιτυχία και παραμένει να είναι ε, επιτυχές νόμισμα. Στο μεταξύ μεσολάβησε η οικονομική κρίση, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ορισμένοι βγήκαν ε, πιο εύκολα από την οικονομική κρίση ή βγαίνουν και άλλοι θα βγουν πιο δύσκολα. Και τώρα καλούμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης να βρούμε τους τρόπους εκείνους και τα μέσα που χρειάζονται για να ξεπεράσουμε την κρίση. Διαπιστώνουμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς στήριξη και διάσωση, όχι επειδή έχει πρόβλημα το ευρώ αυτό καθ' αυτό, αλλά επειδή μεμονωμένε χώρε έχουν προβλήματα να αντιμετωπίσουν το χρέος τους και να εξυπηρετήσουν το χρέος τους προς τις χρηματαγορές και οι χρηματαγορές αρνούνται να τους δώσουν και άλλα χρήματα, να τους δανείσουν. Αυτό είναι ο κίνδυνος, έτσι πρέπει να τον περιγράψουμε, ότι βασικά δεν είναι πρόβλημα των χρηματαγορών αυτό, αλλά είναι πρόβλημα των μεμονωμένων κρατών. Και αυτό το πρόβλημα, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα, θα πρέπει να το λύσουμε στη ρίζα του, στην αιτία του και όχι αλλού. Και αυτό τι σημαίνει. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταξύ άλλων σημαίνει ότι εμείς όλα τα εθνικά κοινοβούλια μαζί θα πρέπει να φροντίσουμε οι χώρες αυτές να δουν την αλληλεγγύη μας, να βγουν από αυτή την κρίσιμη κατάσταση και να μπορούν να δρουν και από μόνες τους. Γιατί ε, αυτοί οι ε, μηχανισμοί είναι για τη διάσωση. Δεν είναι λόγος ε, αυτός σκοπός για τα κράτη. Ακούσαμε ότι το Βέλγιο ξεπέρασε μια δύσκολη κατάσταση ε, με επιτυχία. Γνωρίζουμε και για τη Λετωνία. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα του παρελθόντος επιτυχημένα στα οποία μπορούμε να προσανατολιστούμε. Άλλο τώρα είναι το θέμα της τραπεζικής οικονομίας. Βεβαίω και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίω και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις τράπεζες. Αλλά ερωτώ. Σε σχέση με αυτό που είπε ένας αυστριακός συνάδελφος προηγουμένως. Αυτές τις χρηματαγορές δεν θα πρέπει να τις ρυθμίσουμε. Γιατί εμείς πρέπει να δρούμε πυροσβεστικά και να ε, στρεφόμαστε κατά της διπλανής πυροσβεστικής και λέμε να σβήσει εκείνη περισσότερο. Όχι, να πάμε όλοι μαζί να πιάσουμε τον εμπριστή. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ελεγγύη ακριβώς για τις χρηματαγορές και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν το αντιμετωπίζουμε στη ρίζα του και γεννιούνται και νέα προβλήματα μετά. Ε, Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στους ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έξι παρακαλώ είναι ευρωβουλευτές. Αν θέλετε απαντήσεις προσπαθείτε να μην μακρηγορείτε, όχι πάνω από ένα λεπτό. Ιάννη, παρακαλώ πρώτη κυρία Ποδηματά. Thank uh, Ευχαριστώ πολύ Σάρων. Καταρχάς, συνεχίζοντας από αυτό που σας ρώτησε η κυρία Λούλινγκ προηγουμένως, δεν νομίζω ότι της απαντήσετε και παρόλο που ξεκίνησα από ένα τελείως διαφορετικό σημείο, γιατί εγώ είμαι εισηγήτρια για την καινοτομία στη χρηματοδότηση και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόσο γρήγορα ενέκρινε την πρόταση που έγινε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Σαφής αναφορά στη φόρο στο τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών και έλεγε ότι πρέπει να είναι μια επιλογή που γρήγορα πρέπει να εξεταστεί και σε επίπεδο παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό και σε επίπεδο ευρωζώνης. Και η πρώτη ερώτηση προς τον πρόεδρο Γιούνκερ, πώς ε, προτίθεστε να δώσετε συνέχεια σε αυτό, ότι για πρώτη φορά ε, μπαίνει αυτό στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και δεύτερο, εμπνευσμένη από τη συζήτηση που γίνεται εδώ, αλλά και από ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύουν σήμερα οι Financial Times, θέλω να σας πω τα εξής εκτιμά, αξιολογεί τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τονίζει ότι υπάρχει ένας αόρατος εχθρός και καταπολεμά τις προσπάθειες των Ευρωπαίων ηγετών να αντιμετωπίσουν την κρίση του χρέους. Και αυτός ο αόρατος εχθρός ονομάζεται αυξανόμενος ευρωσκεπτικισμός. Ακούσαμε σχόλια από πολλούς συναδέλφους εθνικών κοινοβουλίων. Τίθεται ένα ζήτημα που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Πώς να εξηγήσω εγώ στους ψηφοφόρους μου το α, το β. Και επίσης λαμβάνοντα υπόψη ότι σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, στην Νότια Ευρώπη, οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι φέρνουν τεράστιο βάρος για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Στη Βόρεια Ευρώπη οι πολίτες και οι φορολογούμενοι έχουν την αίσθηση ότι τους ζητάνε πάλι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν τους λεγόμενους αρματολούς. Αμαρτολούς. Συγγνώμη. Αυτή είναι η πιο ε, επικίνδυνη κατάσταση και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από οποιαδήποτε παραβίαση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Σα ερωτώ αυτό, πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Πιο γρήγοροι να είστε. Parlo in Italiano, così. Θα μιλήσω Ιταλικά, γι' αυτό θα είμαι και γρήγορο. Μια ερώτηση προ τον Επίτροπο Ρεν, λέει ο κύριο Ντομένιτσι. Μια ερώτηση προ τον Επίτροπο Ρεν. Ε, γενική, αλλά αφορά ιδιαίτερα την Ιταλία. Εχθές επαναλάβατε ότι για να αξιολογήσετε ε, τα σχέδια των κυβερνήσεων θα συνυπολογήσετε και ε, το ιδιωτικό χρέος, όχι μόνο το δημόσιο. Αυτό πώς θα γίνει. Πώς θα επηρεάσει τη δυνατότητα μιας ε, χώρας να αποσβέσει το δημόσιο χρέος. Αυτό τι σημαίνει. Στο 120% είναι το δημόσιο χρέος στην Ιταλία. Θεωρείται φερέγγια γιατί είναι πολύ μεγάλη αποταμίευση των οικογενειών και των οικοκυριών. Και τι θα πάρετε τα χρήματα από τους ιδιώτες. Και αν είναι σωστή αυτή η ε, ερμηνεία, πώς θα αντιδράσουν πιστεύετε οι χρηματαγορές. Ευχαριστώ. Το ήξερα ότι μπορούσες να περιοριστείς το ένα λεπτό. Ο κύριος Γκερέρο. Εδώ είμαι κύριε Γιούνκερ, κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το μόνιμο ε, μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή μας εδώ έκανε μια νομοδότηση και ενέκρινε την έκθεση η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων όπου ε, ζητούν ε, εναλλακτικά να επανακαταρτιστεί η πρόταση του Συμβουλίου, να αναδιατυπωθεί ή να γίνει κάποιο είδος δέσμευσης, δήλωσης ότι θα μπουν και κοινοτικά στοιχεία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αλλά και στη λειτουργία αυτού του μηχανισμού σταθερότητας. Στο Κοινοβούλιο θα ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα πριν συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 24 και 25 του μηνό και πιστεύω ότι ο κύριο Γιούνκερ ενέχεται στην όλη αυτή η διαδικασία διαλόγου με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την εξέβρεση λύσεων και τέτοιων ασφαλιστικών δικλείδων. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Βίκυ Φόρτ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα τις απαντήσεις κύριε Γιούγκερ προς την κυρία Λούλινγκ. Ε, ήσασταν σαφέστατος. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σε μεγάλη σύγχυση για το σύμφωνο, γιατί μπορεί αφελώς να πίστευα ότι θα αφορούσε περισσότερο τις τράπεζες. Βλέπουμε διάφορα ερωτηματικά που έχουν οι Moody's για τις ισπανικές τράπεζες. Είδαμε ότι η Ιρλανδική κρίση οφείλεται στις τράπεζες κατά κύριο λόγο και η έλλειψη εμπιστοσύνης πιστεύω και από τα stress test, τα δοκιμές αντοχής, τις περσινές των τραπεζών, χρειάζεται να έχουμε τέτοια τεστ τα οποία να μπορούμε να ε, υπολογίζουμε και να είναι αξιόπιστα. Και από εδώ και πέρα τι γίνεται τώρα. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να χρειαστεί ε, αύξηση του κεφαλαίου των τραπεζών. Τα κράτη-μέλη, ε, λέει, θα πρέπει να Ε, ρυθμίσουν αυτά τα θέματα νομοθετικά. Μα το πρόβλημα δεν ήταν ε, το δίκαιο που ίσχυε για τις πτωχεύσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, ήταν διασυνοριακό. Σήμερα το πρωί κύριο Σόιμπλε είπε ότι κάθε κράτος μέλος συμφώνησε ότι θα σώνει τις τράπεζες εάν έχουν προβλήματα ρευστότητα και κεφαλαίου στα αυτά τα stress test. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε περισσότερο. Ευχαριστώ, Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσα να ακούσω στην αρχή τη παρουσίασή σα. Έχω τι εξή ερωτήσει. Βλέπουμε εδώ ένα αποτέλεσμα που μας δείχνει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τις χώρες αυτές να προσφύγουν στο μηχανισμό. Αλλά είναι πιο σαφής ε, η περιγραφή για το πώς θα προσφύγει στο μηχανισμό παρά τι θα γίνει με το κεφάλαιο και πώς θα στο δώσουν. Ε, δημιουργήθηκε ο μηχανισμός στήριξη στην αρχή για την Ελλάδα, τώρα γίνεται μόνιμος θα συμμετέχει και η ιδιωτική αγορά, αλλά πού είναι το δεύτερο παράρτημα για τις λεπτομέρειες, για τη διάσωση, το bailout κτλ. Τα έχω μπλέξει λίγο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα στην πράξη και στη βάση ομοφωνίας. Δεύτερον, υπάρχουν πολλοί δείκτες εδώ και ταυτόχρονα ε, επεξεργαζόμαστε και νέους δείκτες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Εγώ είμαι και συγγήτρια. Γιατί δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε τα δύο και να τα βάλουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αντί να ελέγχει μία χώρα την άλλη για το πώς θα φτάνει σε ένα στόχο, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς ορίστηκε καν στην αρχή, το τελευταίο για τις τράπεζες. Περιέργως πώς οι χώρες υποτίθεται ότι επεμβαίνουν όταν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα των τραπεζών τους, των ιδίων και υπάρχει και ένα αίτημα οι χώρες να αναπτύξουν δική τους νομοθεσία για τον έλεγχο τραπεζών που πτωχεύουν. Μα όταν μια χώρα είναι σε πτώχευση, ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος. Ε, είναι ενιαίος, αλλά για τις τράπεζες λέτε εθνική νομοθεσία όταν πτωχεύει μια τράπεζα. Μα το Κοινοβούλιο είχε προτείνει ευρωπαϊκή προσέγγιση, όχι εθνική. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα Χίμπνερ. Ευχαριστώ. Η Βίκη με κάλυψε, είχα την πρώτη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω, ομά, τα λεφτά που θα τα βρείτε για την αύξηση κεφαλαίου, ιδιαίτερα ε, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο κεφάλαιο. Και ποτέ δεν ακούσαμε στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Χαίρομαι που σήμερα έρχεται αυτό το θέμα. Ε, και θέλω να ρωτήσω τον Ζαν Κλοντ. Οικονομική διακυβέρνηση λέτε σύμφωνο ευρώ και με διαδικασία και ευκαιρία opt-in για χώρες που δεν είναι χώρες του ευρώ. Και δεν το κάνουμε μόνο επειδή εσύ θες να προεδρεύεις σε μια σύνοδο των 27 υπουργών, αλλά αυτό τώρα πώς θα το οργανώσετε. Ποιος βάζει κανόνες, ε, τα κατόφλια, το benchmarking, πώς θα μπει αυτό στο σύστημα που έχουμε για τις χώρες των 17 ε, του ευρώ ή θα έχουμε άλλη παράλληλη κατηγορία τώρα ξαφνικά. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το διαμορφώσετε αυτό στην πράξη. Ευχαριστώ. Και τα άσχημα νέα τώρα είναι ότι έχετε πέντε λεπτά έκαστος. Είχατε περισσότερο χρόνο προηγουμένως, τώρα πρέπει να επιταχύνετε. Δεν ξέρουμε με ποια σειρά. Κύριε πίτροπε εσείς πρώτος, ποια σειρά θέλετε να απαντήσετε, μια που μιλήσετε τελευταίος, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, Σαρών πολύ δίκαιο και πολύ μεγάλη καλοσύνη σου. Ε, πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις. Δεν θα επιλέξω, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Θα αφήσω και μερικές ερωτήσεις για τον Ζαν Κλοντ και τον Ματόλση, για να ε, κερδίσω χρόνο. Πρώτον, αυτό που ρώτησαν η Βίκη Φόρτ και η Ντανούτα Χίμπνερ για τις τράπεζες. Βίκη, είσαι κάπως αρνητική νομίζω και επιφυλακτική για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα των τραπεζών. Κατά την άποψή μου, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στην αναθεώρηση και μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής του δημοσιονομικού κανονισμού ε, και της εποπτείας. Με δικές σας αποφάσεις όλων των κρατών μελών μετά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγηθήκαμε εκεί σε τρεις επόπτες ε, και για τις τράπεζες και για τις ασφάλειες και για τις securities. Ε, ό,τι αφορά την εποπτεία και ε, τη μακροοικονομική σταθερότητα. Αυτό το συμβούλιο, το e SRB, ε, έχει πρόεδρο τον κύριο Τρισέ της Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί είναι το σημαντικό αυτό. The main η βασική αδυναμία ε, του προηγουμένου γύρου των stress test που έγιναν πέρσι την άνοιξη και το καλοκαίρι στις τράπεζες είναι το εξής. Λόγω έλλειψης ομοιομορφίας και εφαρμογής αυτών των τεστ υπήρξε αυτή η δυναμία. Τώρα το stress test δεν θα αφορά μόνο τις τράπεζες αλλά και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της εποπτείας και της χρηματοοικονομικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Θα αποφασίσει ε, λοιπόν η αρχή για τις τράπεζες για την κοινή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθεί και στα 27 κράτη-μέλη και θα γίνουν και τα stress tests. Και μόλις θα έχει γίνει αυτό, οι δοκιμές φυσικά θα ολοκληρωθούν μέσα στον Μάρτιο, Απρίλιο, άντε και Μάιο. Θα γίνει μετά μια αξιολόγηση όλων και πριν το καλοκαίρι αυτά τα τεστ θα δημοσιευθούν. Μέχρι τότε είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα έχουν τέτοιες ρυθμίσεις κάνει ώστε να μπορεί να γίνει παράλληλα αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι λοιπόν η αγορά. Φυσικά είναι καλύτερο να έχουμε τη χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές. Αν αυτό δεν αρκέσει, δεύτερη γραμμή άμυνας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν εθνικές ε, οικονομικές αντιστάσεις ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη κεφαλαιοποίηση. Τώρα, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, όπω το EFSF, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενό προγράμματο για μια χώρα και όχι χωριστά. Γι' αυτό και το μέσο αυτό ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ιρλανδίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτές, ή, ε, αυτά τα stress test να γίνουν με ομοιομορφία Και όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό παράλληλα να μπορούμε να χειριστούμε τις συνέπειες των πληροφοριών που λαμβάνουμε για αυτά τα stress test. Έπειτα, πριν να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι υπήρξε μια ανάμεση ερώτηση για το ιδιωτικό χρέος σε σχέση με την Ιταλία. Ε, μία από τις καινοτομίες και τις αποφάσεις κλειδιά σήμερα στο Συμβούλιο Κοφίν και φαντάζομαι και στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα θα είναι να εγκριθεί η εισαγωγή ε, του κριτηρίου του χρέους στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με σοβαρό τρόπο. Ίσως θα θυμάστε ότι στη συνθήκη και στο Σύμφωνο το έλλειμμα και το χρέος είναι ίσα όσον αφορά το βάρος τους. Για κάποιο λόγο όμως μόνο το έλλειμμα θεωρήθηκε μεταβλητή στην εκτίμηση της οικονομικής πολιτικής. Τώρα πρέπει όμως αυτό να διορθωθεί και είμαι πολύ ικανοποιημένο ε, για το ότι το κριτήριο ε, αυτό του χρέους θα γίνει σοβαρό κριτήριο με ετήσια έκθεση για την μείωση του χρέους. Και σε αυτό το πλαίσιο κάναμε τον συμβιβασμό ότι σχετικοί και μεταβλητέ όπω το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέο, από τη στιγμή που έχει αντίκτυπο στι δυνατότητε τη χώρα να εξυπηρετήσουν το δημόσιο του χρέος το δημόσιο τη χρέο, θα ληφθεί υπόψη. Και είναι λογικό αυτό κατά τη γνώμη μου. Τέλο, χρησιμοποιήσω το τελευταίο μου λεπτό για να πω. Η κυρία Φερέιρα αναφέρθηκε σε δείκτες που είναι πολύ σημαντική για το δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης και των μακροοικονομικών ανισορροπιών και Πόσο γνωρίζω, η συζήτηση για αυτό το θέμα για κάποια κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη τη χώρα μου είναι η εξή, ότι δεν σημαίνει και ποτέ δεν θα σημάνει ότι θέλουμε να αποδυναμώσουμε τις εξαγωγέ οποιοδήποτε χώρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξωπραγματικό, εξωγήινο. Θα ήταν ε, ε, ε, έω και βλακώδη συμπεριφορά και σίγουρα δεν είναι δική μα πρόθεση. Η πρόθεσή μας είναι να εξετάσουμε τι ιδιαίτερα στις χώρες τις ελληματικές, γιατί εκεί είναι οι πιο πιεστικές ανάγκες να διορθωθεί δηλαδή η ανταγωνιστικότητα, αλλά επίσης και στις πλονασματικές χώρες να δούμε ποιες, ποια μέσα υπάρχουν για τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις και για να αυξηθεί η εγχώρια ζήτηση. Θα έλεγα ότι είναι κάπως... Ε, η Μπάγερ Μούνχεν να παίζει κόντρα στην Μιλάν ε, ε, σήμερα. Δεν θέλουμε να, να ισοπεδώσουμε το παιχνίδι, ζητώντας από την Bayern Μίνχεν να παίξει διαφορετικά. Όχι, θέλουμε να συνδυάσουμε τις, την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα και έτσι να δημιουργήσουμε δυνατότητες και προϋποθέσεις για μια καλύτερη γενική απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ο στόχος ε, της διαδικασίας αυτής ε, και έτσι σκοπεύουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω... Ζαν ε, Κλόντ, ότι θα πρέπει να μείνει στα πέντε λεπτά. Μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για τα Eurobond. νομίζω ότι έχουμε πει ήδη αρκετά. διαπιστώνουμε ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και τα νέα μέσα που δημιουργούμε μετά από λίγο χρόνο θα πρέπει να τα συγκρίνουμε με το τι θα ίσχυε αν είχαμε εισαγάγει ευρωομόλογα. Αν το δούμε εκ των υστέρων και το συγκρίνουμε, Ε, θα δούμε ότι είναι μηδεμινές οι διαφορές και ότι θα ήταν πιο εύκολο να λειτουργήσουμε με βρομόλογα αλλά αυτό θα το πει το μέλλον. Για τα CDS δεν λέω τίποτα, ε, γιατί δεν έχω χρόνο. Για τις συλλογικές συμβάσεις, αυτό που είπα δεν ήταν καθόλου ηρωνικό. Το είπα σοβαρά και εγώ γνωρίζω ότι στο τοπίο των συλλογικών ε, συμβάσεων και στις διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να γνωρίζουν όλοι τι γίνεται. Αν ζητούμε όμως άτα και στην Ευρώπη ολόκληρη ε, αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ε, το θεωρώ σοβαρό αρκετά για να το αναφέρω και το συζητάω. Δεν ήταν καθόλου ηρωνικό. Και επίσης, δεν είπα εγώ ότι θα πρέπει να βρούμε κάπου το κεφάλαιο. Το ανέφερα, το χαρακτήρισα callable capital, δηλαδή ένα κεφάλαιο που μπορεί να κινητοποιείται. Δηλαδή έχουμε ένα κεφάλαιο το οποίο έχει καταβληθεί, υπάρχει, ένα άλλο κεφάλαιο ε, που μπορούμε να το βρούμε, να το κινητοποιούμε, πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που θα είναι πραγματικά καταβληθέν και για κάποιες εγγύησεις. Αυτά όμως θα το δείξουν οι συζητήσεις των επομένων εβδομάδων. Για το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Εγώ καταρχήν είμαι υπέρ παρόλο που γνωρίζω ότι για λόγους ε, δεοντολογικούς και ηθικούς πάντα συμφωνούμε, αλλά εγώ είμαι υπέρ και για λόγους δικαιοσύνης, όχι μόνο ηθικοπλαστικούς. Και επειδή ε, με ενοχλεί πάρα πολύ, παρόλο που δεν έχει άμεση σχέση αυτό επί της ουσίας, το γεγονός ότι ε, στον χρηματοπιστωτικό κόσμο συμβαίνουν πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα θεωρούσα ότι θα επαναλαμβανόντουσαν ε, ε, ε, μετά την κρίση. Αυτά τα μπόνους που οργιάζουν. Πώς να εξηγήσουμε και εμείς στον κόσμο αυτά που κάνουμε. Γιατί ο κόσμος ρωτάει, τι κάνετε για τα μπόνους. Γιατί σώνετε τις τράπεζες παρόλο που δεν σώσαμε μόνο τις τράπεζες και, και μετά μας λένε τι σώνεται και μετά αυτές οι διεθνείς τράπεζες σωρεύουν τέτοιο κεφάλαιο και πληρώνουν τόσο τεράστια μπόνους. Και έρχεται ολόκληρη η πολιτική τάξη να εξηγεί προβλήματα για τα οποία δεν αφήνεται η ίδια η πολιτική. Και ευθύνονται αυτοί οι τρομεροί κερδοσκόποι που απομιζούν το σύστημα. Και θεωρώ πάρα πολύ ότι βεβαίω θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα των πόνου, να το ρυθμίσουμε και με τρόπο μαζικό και συνολικό. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να πολιτευόμαστε και να εξηγούμε τι κάνουμε στον κόσμο. Για το τέλος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών το συμφωνήσαμε. Δεν ήταν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συμφωνήσαμε να το μελετήσουμε Explore και develop είναι ο όρος. Θα το διερευνήσουμε και θα το αναπτύσσουμε στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Θα πρέπει να συνεχθούμε όμως με ποια βάση μετρήσιμη θα γίνει αυτό, ε, σε τι θα επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα. Πώς θα γίνει αυτό, ή μόνο στον κίνδυνο, ή προϊόντα που συνδέονται και συναλλαγές που συνδέονται με ρίσκο. Όλα αυτά θέλουν μελέτη και θα χρειαστούν και χρόνο. Και όταν ρυθμίσουμε το κάθε θέμα ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε και γέφυρες και προς άλλους εκτός Ευρωζώνης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, περιμένουμε προτάσεις τώρα που πρέπει να γίνουν. Εγώ έχω και μια αλλεργία απέναντι στην ιδέα που χωρίζουμε τις χώρες σε βορρά-νότο, οι τη βόρη, η αμαρτωλή νότη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι πάνε έτσι οι διαχωρισμοί και οι γραμμές θα πρέπει να μάθουμε με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα να μην κάνουμε σφάλματα στα οποία είχαμε πέσει στο παρελθόν. Παρόλο που πρέπει να πω ότι αν δεν υπήρχε λύση, αν δεν λυθούν τα προβλήματα των λεγόμενων νοτίων κρατών, θα τους βγει πιο ακριβά των βορείων. Ε, παρά αυτό που κάνουμε τώρα και ε, ε, ψάχνουμε λύση με τους φίλους μας ε, της ε, περιφέρειας, γιατί είναι πολλές οι τράπεζες από τον ενάρετο βορρά που θα εκπλαγεί κανείς ε, εάν συμφωνούσαμε να αφήσουμε στη μοίρα τους τις χώρες αυτές. Χώρες του ευρώ και χώρες εκτός ευρώ μπορούν, δεν θα πω να προσχωρήσουν στο σύμφωνο για το ευρώ, γιατί είναι βαριά κουβέντα, αλλά αυτές οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο ευρώ, ε, στα προγράμματα σύγκλησης τους και στα εθνικά τους προγράμματα έχουν στόχους ε, και θέλουν να δανειστούν στόχους από το πρόγραμμα, από το σύμφωνο του ευρώ και να τους εφαρμόσουν στη χώρα τους, τότε είναι ευπρόσδεκτα ε, όλα τα κράτη και τα 27 κράτη μπορούν να δρουν με τον ίδιο τρόπο και θα πρέπει να λογοδοτούν. Μίλησε έξι λεπτά και έξι δεύτερα, παρακαλώ. Ναι. έχασες, όμως έχεις έλλειμμα, γιατί είπα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επανέλθω στο παρατήρηση του Γερμανού συναδέλφου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι η κρίση του ευρώ, της ευρωζώνης. Είναι ένα σύνολο οικονομικών προβλημάτων ορισμένων μεμονωμένων χωρών. Αυτό είναι το ζουμί της συζήτησής μας, ε, γιατί η συζήτηση αφορούσε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για ε, το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Γιατί κάτω από το ευρωπαϊκό εξάμενο έχουμε εθνικά προγράμματα ή ατομικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα καταλήξουν σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, με ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη οικονομία. Αυτή, αυτό είναι το ζουμί αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Ε, τώρα δίνω το λόγο στον Σύμπροεδρο που χρειάστηκε να κάτσει εδώ δίπλα μου και να ελέγχει το χρόνο ομιλίας του καθενός. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. να κάνω μία παρατήρηση καταληκτικά. Ξεκίνησα σήμερα λέγοντας ότι στις 15 Μαρτίου το 1848 έγινε μια επανάσταση στη Βουδαπέστη που πέρασε από την πέστη στη Βούδα από μία γέφυρα Τότε υπήρχε μόνο μία γέφυρα. Πέρασε ο κόσμος από αυτή τη μία. Τώρα έχουμε δέκα. Δέκα και αυτή η παλιά ανακαινίστηκε. Πρόσφατα. Οι γέφυρες είναι λοιπόν το θέμα. Όχι μόνο στη Βουδαπέστη, αλλά στην Ευρώπη γέφυρες που διανύει κανείς με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, με, το, με ένα λεωφορείο. Οι γέφυρες είναι αυτές που μας συνδέουν. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη και ισχυρότερη Ευρώπη και καλύτερη ζωή να έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια γέφυρα που πρέπει να φτιάξουμε και να χρησιμοποιήσουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να κλείσουμε λέγοντας ότι εδώ υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός ανάμεσα στα διάφορα μέσα. Αν είναι πρώτο και καλύτερο το σύμφωνο για το ευρώ, το εξάμενο φυσικά δημιουργεί ένα καλό γενικό πλαίσιο, αλλά θα ήταν καλό να πούμε ότι η φιλοδοξία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε κάποιο βαθμό το πακέτο των έξι μέτρων να μπει ως προτεραιότητα, γιατί εκεί περιλαμβάνονται νομοθετικές δεσμεύσεις και προβλέπουμε να βάλουμε και αν μάλλον φτιάξουμε αυτό το πακέτο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και τη σύνδεση με την εποπτεία και με, το πλαίσιο, και με διάφορα άλλα εργαλεία. Αυτή θα παραμείνει λοιπόν η δική μας ε, φιλοδοξία και ελπίζουμε πως θα έχουμε κάτι πιο συντονισμένο στο τέλος. Να σας θυμίσω τέλος ότι υπάρχει μια άλλη διακοινοβουλευτική συνάντηση που διοργανώνεται από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δημοσιονομικά θέματα και τη συνεργασία ανάμεσα, τη σχέση ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τους εθνικούς ε, προϋπολογισμού στο πλαίσιο του, εξαμήνου, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αυτή διοργανώνεται για τις 20, 13. 13 Απριλίου του 2011. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι και σημειώστε παρακαλώ αυτή την επόμενη συνάντηση. Να ευχαριστήσω και τους ομιλητές μας ε, για το ανοιχτό τους πνεύμα, γιατί με ανέχθηκαν που τους μάλλον για το χρόνο πέρα της συνεδρίασης.